Non, elle n'est pas là. Aujourd'hui, il faudra se contenter de, de son vice-président. Bien. Κυρίε και κύριοι, εάν δεν έχετε αντίρρηση να ξεκινήσουμε το σχέδιο μέσης διάταξης ε, δεν δημιουργεί κάποιο, κάποια δυσκολία. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στην έγκριση των πρακτικών τη προηγούμενη συνεδρία. Υπάρχουν σχόλια από αυτού. Εάν δεν υπάρχουν, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Κάποιες ανακοινώσει του Προέδρου. Το πρώτο είναι σημαντικό νομίζω. Οι διαπραγματεύσει ε, τον τρίλογο ό,τι αφορά την, τον μηχανισμό διασύνδεση στην Ευρώπη ολοκληρώθηκε ευτυχώ τη νύχτα ε, τη 17η Μαρτίου το κείμενο αυτό που ανακρίθηκε από το Συμβούλιο έκτοτε θα αποτελέσει αντικείμενο επιστολής επιβεβαίωσης 19 Μαρτίου να ευχαριστήσω την ομάδα των μεταφορών τον κύριο Μαρινέσκου, τον κύριο Τεντίτσκα ε, και όσους ε, συνεισέφεραν για να ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση εσίως Βεβαίω θα πάρθουν κάποιε αποφάσεις αργότερα σε ό,τι αφορά τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία, όπως όλα τα δημοσιονομικά ζητήματα. Φτάσαμε όμω σε ένα ικανοποιητικό και λειτουργικό συμβιβασμό. Οι, οι, οι επιτροπές Τρέν, Ήτρε ε, θα ψηφίσουν στι 25 Μαρτίου πριν την Ολομέλεια, στην πρώτη ανάγνωση, θα ψηφιστεί και θα έχουμε ολοκληρώσει έτσι και τον, αυτόν τον την τις βγαίνουν αυτό σε πολύ σημαντικό μηχανισμό. Πριν ξεκινήσουμε την ακρόαση για τις ε, ποταμιώσεις οδούς, ε, θέλω να καλωσορίσω μια ομάδα από τη Σάξεν Άνχαλτ ε, που τους έχει καλέσει ο κύριος Ντίτερ Χολ. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι ο ίδιος επ' αυτού. Αγαπητοί φίλοι, ε, περάσαμε μέσα από την Έση, ήρθαμε όμως από την ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας έχουμε εδώ κοντά μας σήμερα. Εντάξει λοιπόν, καλωσορίζουμε και τον κύριο Κρίς Φιλτσέπε, τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής Δημοσίων Μεταφορών, ε, Πατών Δημοσίων Μεταφορών του Βερολίνου, τους οποίους, τον οποίο έχει καλέσει ο πρόεδρος ε, Μάικλ Κράμερ. Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, θα έχετε λάβει, θα βρήκατε μπροστά σας την, το, την έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Μεταφορών 160 σελίδες. Αυτό δείχνει έτσι με πόση, ε, πόση αυτοαπάρνηση εργάστηκαν Εργαστική Επιτροπή αυτή. Ευχαριστώ και την Γραμματεία ε, για τη δουλειά αυτή, την άχαρη δουλειά, η οποία όμω είναι και χρήσιμη, διότι έτσι θα μπορούν και οι βουλευτέ να λογοδοτήσουν στι υποψήφιό του ε, στο τέλο τη εντολή του, στα πλαίσια τη ε, μελλοντική του ε, εκλογική εκστρατεία ενδεχομένω. Μια απόδειξη ότι η Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δουλεύει για του πολίτε. Το έργο τη Επιτροπή μα έχει ω απότατο στόχο να βελτιώσει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας στον τομέα των μεταφορών. Ε, το τομέα των μεταφορών άλλωστε είναι ένα τομέα ε, που επηρεάζει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Να ευχαριστήσω τους ε, βοηθούς μας, τους συμβούλους μας που μας βοήθησαν, μας έσπρωξαν, ορισμένε φορέ μα μαστίγωσαν κιόλα σε αυτή την πενταετία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να είμαστε έτσι παραγωγικοί. Θα υπάρξει και μια ψηφιακή εκδοχή του κειμένου στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Μεταφορών. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο κεντρικό ζήτημα. Ένα ζήτημα που με απασχολεί ιδιαίτερα. Οι εσωτερικές πλωτές οδοί στα πλαίσια της ε, ε, διαδικής ε, μεταφοράς. Ε, ξέρετε ότι υπάρχει η Λευκή Βίβλος του 2011 ε, που περιλαμβάνει ένα οδικό χάρτη έτσι ώστε έως το 2030 να φτάσουμε σε 30% σε ό,τι φορά τη μεταφορά των εμπορευμάτων ε, μακράς, μεγάλων αποστάσεων Θέλουμε να περάσουμε βεβαίως σιγά σιγά προς το σιδηρόδρομο, αλλά και οι πλωτές οδοί είναι ένα σημαντικό παράγοντα. Ο στόχο είναι το 2050 να φτάσουμε στο 50% ε, των μεταφορών αυτών. Ε, ξέρουμε ότι ε, δεν είναι σωστή η κατανομή δεν είναι, τόσο ισομερή η κατανομή για ιστορικού λόγου ορισμένε φορέ. Κάποιε χώρε πάντω είναι πολύ προχωρημένε. Η κατοχώρη, παραδείγματο χάρη, ο Βίλμερ Λενκόμπ, εδώ, τον οποίο χαιρετίζω, είναι στην πρώτη ε, γραμμή. Είναι η, πρώτη, πάνω από 30% ήδη. Έχετε περάσει, το έχετε φτάσει πολύ πριν το 2030 αυτό. Και το 2050 θα το. Θα το στόχο του 2050 μάλλον αρκετά σύντομα. Γνωρίζουμε ότι αυτή η μεταφορά ε, προς το ποταμί εισοδούς ε, έχει πολλά θετικά στοιχεία όχι μόνο για το κλίμα και το περιβάλλον αλλά και σε ό,τι αφορά την ε, αποτελεσματικότητα. Δίνονται, υπάρχουν πολλές δυνατότητε σε αυτή τη συγκεκριμένη τον τρόπο μεταφοράς και υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης. όπως ε, για τις θαλάσσιες οδούς ε, θα πρέπει και για τις ποταμίσιες οδούς ε, να μπορέσουμε να περάσουμε σε άλλα καύσιμα πέρα από τον ντίζελ, έτσι. Έχουμε εδώ μαζί μας τέσσερις εμπειρογνώμονες. Θα τους ακούσουμε διαδοχικά. Την κυρία Καρίνη Σέπερ πρώτα, που είναι η διευθύντρια του Europe του Map Navigation Europe, ο κύριος Ντόραφτσικ, ο οποίος είναι ε, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ναυτιλίας, ο κύριος Έρικ Σούλτς, αντιπρόεδρος του König Nature Weil και άλλος ένας ομιλητής. Θα έχει το καθένας το λόγο για 6 λεπτά. Ξέρετε ότι είναι συγκεκριμένο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην κυρία Κοπτσίνκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει και αυτή πέντε λεπτά στη διάθεσή της ε, για να ξεκινήσει την συζήτηση αυτή. Κυρία Κοπτσίνκα, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε για το λόγο. Θέλω να υποσχεθώ ότι θα προσπαθήσω να σεβαστώ το χρόνο που μου έχετε δώσει. Συνήθως δεν το πράττω αυτό. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή που οργανώσε αυτή την ακρόαση και που εξέτασε τα τελευταία πέντε έτη αυτό το πολύ σημαντικό κλάδο. Πρόκειται για ένα τομέα της οποίας η σημασία να γνωρίζεται από όλους. Όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας για τις προσπάθειες να αντιμετωπίσετε τη δυναμική αυτού του συγκεκριμένου κλάδου. Καταρχήν, έχοντας καταθέσει και ψηφίζοντας ε, το ψήφισμα που καλεί για ένα πρόγραμμα follow-up, ένα πολύ επιτυχές πλαίσιο για να υποστηρίξουμε τις εσωτερικές πλωτές οδούς και επίσης ε, για τη σαφή έκκληση για χρηματοοικονομική υποστήριξη για την εφαρμογή του προγράμματος. Το ψήφισμα θα υποστηρίξει τα συμπεράσματα τη ενδιάμεση έκθεση πρόοδρου ΝΑΙΑΔΕΣ 2 και την έκθεση για τι ε, ποτάμιες μεταφορές. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια σε πάρα πολλές περιπτώσεις η Επιτροπή Τραν ε, αναγνώρισε τη σημασία του κλάδου της ε, εσωτερικής ναυσιπλοείας. Αναφέρεστε πάρα πολύ σε φως στον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι εσωτερικές πλωτές οδοί, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στο θέμα των διατροπικών μεταφορών κτλ. Για τις εσωτερικές πλωτές οδούς νομίζω ότι όποιο θέμα είχε στην μισή διάταξη τα πέντε έτη επενδύσεις, καινοτομία, μίσου του άνθρακα και κοινωνική διάσταση τα γνωρίζει ο κλάδος και έχει εργαστεί όλους σε όλα αυτά τα θέματα διασφαλίζοντας ε, πως ε, ό,τι και να γίνει ε, θα έχει εγγραφεί στις συνολικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφορές, αλλά και όχι μόνο. Επίσης, Ελπίζω να υπάρξει αναγνώριση ότι η Κομισιόν έχει πάρει πολύ σοβαρά την στήριξη για τον τομέα στο παρελθόν. Επί του παρόντος, να αναφερθώ στο τι υπάρχει επιτάπητο σε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ανάγκη να εφαρμόσουμε τι οδηγίε για τα τεχνικά πρότυπα και για τα επαγγελματικά προσόντα. Και πάλι είναι ένα κλάδο που Επιτροπή Μεταφορών Σημείωσα μεγάλη επιτυχία ε, σε ό,τι αφορά τις συζητήσει για τη σχετική οδηγία για τα προσόντα και χαίρομαι που βλέπω την εισηγήτρια εδώ γιατί μπόρεσε να ξεμπλοκάρει πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις για αυτό το νομοθέτημα. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τα σχέδια καινοτομία για τις διατροπικές μεταφορές, για το πρασίνισμα του στόλου. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε τον τομέα και να σχετίζεται αυτό με όλη την αλυσίδα επιμελητίας. Ε, και επίσης, ε, ε, ακόμη και δεν αμφισβητείται η περιβαλλοντική πτυχή του κλάδου πρέπει να διασφαλίσουμε πώς ο στόλος θα γίνει ακόμη πιο πράσινος και πώς θα ανταποκρίνεται περισσότερο στις ε, προκλήσεις που τίθεται και τις περιβαλλοντικές και σε ό,τι αφορά ε, την ε, κλιματική αλλαγή αλλά και την ποιότητα του αέρα. Επίσης πρέπει να συνεχίσουμε να προσπάθειες να ολοκληρωθεί το δίκτυο TEN-T πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές για τις εσωτερικές πλωτές οδούς το Κοινοβούλιο κάλεσε να υπάρξει περιττέρω χρηματοοικονομική ενίσχυση μέσω του ε, προγράμματος Horizon Ευρώπη. Αυτό προωθήθηκε από την Κομισιόν και το καταθέσαμε στο τραπέζι όταν ε, παρουσιάσαμε και τις προτάσεις μας. Τώρα είναι υπολοκλήρωση μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα των συζητήσεων θα ωφελήσει τον κλάδο και ιδίω ίσως μπορεί να υπάρξει πιθανή αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης υπό το μηχανισμό συνδέοντας ε, την Ευρώπη για τις υποδομές ε, στις εσωτερικές πλούτε οδούς. Και είμαι πεπισμένη ότι δεν, αν και δεν μπορούν να ληφθούν πολιτικέ δεσμεύσει, ότι το αίτημα τη Επιτροπή Τραν για ένα πρόγραμμα ε, συνέχιση ε, στον ΑΙΑΔΕΣ 2 θα εξεταστεί πολύ προσεκτικά όταν θα αναλάβει η νέα Κομισιόν η ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, από τις Ναϊάδες ε, ε, ξεκίνησε ήδη να αναλύει το περιεχόμενο του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου και του προτινόμενου φόλου από τους τελευταίους μήνες. Και πάλι θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση, δυνατότητα να απευθυνθεί σε εσάς ο κλάδος σήμερα και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα ακούσουμε πάρα πολύ προσεκτικά τις δηλώσεις των εκπροσώπων του κλάδου και τις ερωτήσεις που θα θέσουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συμπεριληφθούν και στο δικό μας προβληματισμό για το μέλλον των ευρωπαϊκών πολιτικών για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ε, που υπάρχουν στις εσωτερικές οδούς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια. Κυρία Κοψίνκα, τα καταφέρατε εντός χρόνου. Σας ευχαριστούμε που παρουσιάσατε και τους εμπειρογνώμονες για να μην χάνουμε χρόνο και θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Ντεσέπερ η οποία είναι η διευθύντρια του Inland Navigation Europe. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτές κυρίες και κύριοι. Είναι πάντοτε χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή σας για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, τις εσωτερικές πρώτες οδούς ε, έχετε πάντοτε μια επικοδομητική στάση, χρήσιμη για τη διαμόρφωση της πολιτικής για τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Σήμερα θα σας δώσω κάποια παραδείγματα για τις βιώσιμες εσωτερικές μεταφορές μέσω εσωτερικής ναυσιπλοΐας, όπως ακούσαμε ήδη και από την Κομισιόν. Ε, από άποψη πολυτροπικότητας ε, θα ε, σας περιγράψω και λίγο ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον. Δεν γνωρίζουμε, όπως και εσείς, ε, τι μα επιφυλάσσει το μέλλον. Υπάρχουν κάποιε αβεβαιότητες ακόμη, ωστόσο γνωρίζουμε ποιε είναι οι προκλήσει που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι κοινέ οι προκλήσει αυτέ. Πρέπει να καθασίσουμε τι πόλει μα προσβάσιμες με υψηλό επίπεδο ζωής, ε, γιατί ε, μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει στις πόλεις. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις εκπομπές άνθρακα, τι κλιματικές αλλαγές, σημαντικό για το μέλλον των ε, παιδιών μας. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερο οι εσωτερικές πλωτέ οδοί και να ενταχθούν ε, στην, ε, στο πλαίσιο της κλιματικής πολιτικής συνολικά οι μεταφορές μας. Για το πώς μπορούμε να καταστήσουμε τις, τις πόλεις μας πιο υγιείς και πιο προσβάσιμες. Ξέρετε ότι πολλές από τις πόλεις μας για ιστορικούς λόγους χτίστηκαν πάνω σε ποτάμια. Και αν δείτε σήμερα οι μεγαλύτερες εμπορευματικές μεταφορές αφορούν ακόμα τα οικοδομικά ε, υλικά. Πέρα από τα, τις μεγάλες μεταφορές με τα μεγάλα φορτία λοιπόν υπάρχει, υπάρχουν και υβριδικά πλοία πλέον, δέματα, εμπαρευματοκιβώτια, ε, καθαρά λεωφορεία, υδάτινα ε, και οι πόλεις δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για όλα αυτά Ωστόσο, πρέπει να συνδεθούν οι εσωτερικέ πλωτέ με του άλλου τρόπου μεταφορών και αυτό χρειάζεται χώρο. Χώρο μέσα στι πόλει και εδώ πρέπει να σκεφτούμε πώ ακριβώ θα αξιοποιήσουμε τον υπάρχοντα χώρο από κοινού για, όλες τις, για όλα τα είδη μεταφορών. Επίσης, υπάρχουν πλέον τα πρώτα ηλεκτρικά πλοία, κάποια κινούνται με υδρογόνο, κάποια είναι υβριδικά, έχουμε και ε, ε, συστήματα ε, λιμένων τα οποία επίσης τίθενται σε λειτουργία. Έχουμε όμως και αρκετές προκλήσεις μπροστά μας. Για την ανάπτυξη στο μέλλον χρειάζεται οπωσδήποτε να μειωθεί το κόστος αυτών των τεχνολογιών. Πρέπει να τους δώσουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική ε, για μεγάλες αποστάσεις επίσης, όχι μόνο για τις μικρές αποστάσεις. Και εδώ πραγματικά χρειαζόμαστε να εντάξουμε αυτά τα θέματα στο πλαίσιο και του ΣΕΦ και του Ορίζοντα 2000 Ευρώπη. πώς θα καταστήσουμε εύκολα στη χρήση τις εσωτερικές ε, πλωτές οδούς. Χρειάζεται ψηφιοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και πραγματικά εργαζόμαστε σκληρά για το πώς θα μπορέσουμε να ε, εντάξουμε τις εσωτερικές πλωτές ε, οδούς με την νέα αντίληψη για τη συνδεδεμένη ναυσιπλοεία. Θέλουμε να προσαρμοστούμε στις νέες ανάγκες, αλλά χρειάζεται βεβαίως γρήγορα να προχωρήσουμε και στην ε, αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ε, ναυσιπλοείας. Ηλεκτρονικά έγγραφα, έξυπνες υποδομές για τη διαχείριση κυκλοφορίας, ακόμη και διασυνοριακής, ε, αυτόνομη ναυσιπλοεία, ε, υδάτινα drones επίσης χρησιμοποιούμε. Όλα αυτά θέλουμε να τα εντάξουμε ακόμη περισσότερο στις πολυτροπικές μεταφορές, να συνδεθούν όλες, όλα τα είδη μεταφορών. Όλα αυτά χρειάζονται βεβαίως και αντίστοιχες προσπάθειες και στις μεταφορές και στην ε, εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά για να ολοκληρωθούν αυτά πρέπει να ενταχθούν αυτές οι διαδικασίες και στα προγράμματα ορίζοντα 2000, ε, Ευρώπη και χρειάζεται βεβαίως να καταρτιστούν προδιαγραφές, πρότυπα, να καταρτιστούν ε, ευθύνες, αρμοδιότητες. Επίσης, θα θυμάστε πέρσι το καλοκαίρι το, τη χαμηλή στάθμη των υδάτων αλλά και τις καταστροφικές πλημμύρες που έγιναν στην Ιταλία και σε άλλες χώρες που επηρέασαν ολόκληρο το σύστημα των μεταφορών. Αλλά όχι μόνο τις μεταφορές αλλά και τις ίδιες τις ζωές των ε, πολλών πολιτών. Ε, αυτές οι επιπτώσεις βεβαίως, αυτά τα φαινόμενα μάλλον δεν είναι εξαιρέσεις περιμένουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής να πολλαπλασιαστούν τέτοια φαινόμενα. Όταν λοιπόν εργαζόμαστε επί έργων στην εσωτερική ναυσιπλοεία, ε, να ξέρετε ότι αυτά τα έργα είναι πάντοτε πολυσχηδή και λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από διαστάσεις όπως είναι η βιοπικιλότητα, η κλιματική αλλαγή, η ποιότητα του νερού, η ποιότητα του νερού ως πόσιμου ή ως νερού άρδευσης Πραγματικά η προσέγγιση μας είναι διατομεακή και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τα ευρωπαϊκά προγράμματα να μην ε, χαρακτηρίζονται από ε, κατακαιρματισμό, να μην σκέφτεται ο καθένας δηλαδή το δικό του χωραφάκι, αλλά πώς θα αυτό είναι το σημαντικό, πώς θα μπορέσουμε όλοι μαζί να επενδύσουμε και να ερευνήσουμε και να αξιοποιήσουμε τα πολλαπλά ωφέλη Θέλουμε λοιπόν να έχουμε εσωτερική ναυσιπλοεία, η οποία θα είναι ανθεκτική στο μέλλον, που θα είναι κατάλληλη για τις μελλοντικέ ανάγκες και θέλουμε 50% ε, συγχρηματοδότηση από το ΣΕΦ 2, ακριβώς για να καταστήσουμε την εσωτερική ναυσιπλοεία ανθεκτική στο μέλλον, έτοιμη για το μέλλον ε, και έναντι της ε, ε, κλιματικής αλλαγής και στο ορίζοντας Ευρώπη πραγματικά θέλουμε να σας ζητήσουμε να διατηρήσετε αυτό το, αυτό το δίπολο της, ε, των μεταφορών του κλίματος και της ενέργειας από την άλλη μεριά. Γιατί πραγματικά πρέπει όλες οι δράσεις μας να λαμβάνουν υπόψη και τις δύο διαστάσεις. Ε, Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λίγο στον κύριο Ντουρατσίκ, ο οποίος ε, προέρχεται από το Πανεπιστήμιο του Τσέτσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, θέλω να υπογραμμίσω το γεγονό πρώτα απ' όλα ότι στον τομέα των μεταφορών ε, των θαλάσσιων είναι ένα τομέα ο οποίο είναι ελπιδοφόρος, είναι καινοτόμος, ε, έχει το μέλλον μπροστά του. Και όταν μιλάμε για καινοτομία, ε, υπάρχουν οι πληροφορίες, ε, τα συστήματα στα υπηρεσίες πληροφοριών, στους ποταμούς. Όταν μιλάμε για εσωτερική ναυσιπλοεία, μιλάμε και για ψηφιοποίηση των εγγράφων, για νέες βάσεις δεδομένων. Και αυτά είναι χαρακτηριστικά καινούρια. Οι δεξιότητες ε, των ανθρώπων που προέρχονται στον τομέα αυτών, όλα αυτά αφορούν το μέλλον. Πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα και στις ε, διοικήσεις και στις επιχειρήσεις. Πρέπει να πω ότι η πρώτη υπηρεσία την οποία παρήσχαμε στον τομέα της εσωτερικής ε, νοσηπλοείας έχει να κάνει με τη διαχείριση των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοείας. Θέλουμε να έχουμε μια είναι καλύτερη χρήση των ροών εμπορικών, των εμπορικών ροών, καλύτερη διαχείρισή τους μάλλον, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Εφαρμόστηκε στο νομοθετική πράξη του 2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υποχρεώνει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα όταν έχει επίπεδο νερού κατηγορίας 4 υψηλότερης. Εδώ έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ε, για τους ε, πλειοκτήτες, για τη διοίκηση, για τους πλοίαρχους. Ε, τέσσερις πολύ βασικές υπηρεσίες ε, του συστήματος αυτού βοηθούν να έχουμε μια καλύτερη λειτουργία του συστήματος. Βλέπετε λοιπόν τέσσερα από αυτά, τα πιο σημαντικά. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι το VTT, Vessel Tracking and Tracing, αυτό σημαίνει παρακολούθηση της κυκλοφορίας στα εσωτερικά ύδατα. Το δεύτερο είναι η Προ προς τους πλοιάρχους, προς τους ε, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα, βρίσκεται η θαλάσσια οδός, η εσωτερική, θαλάσσια οδός. Μετά έχουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα ε, μάλλον είναι κάποιοι χάρτες ηλεκτρονικής ε, ναυσιπλοείας και επίσης μια υπηρεσία η οποία ε, επιτρέπει να έχουμε καλύτερες εκθέσεις, ηλεκτρονικές εκθέσεις ό,τι αφορά ε, την πορεία του πλοίου και είναι κάτι που να χρήσουμε και σε επίπεδο υποδομών. Εάν δούμε τώρα τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΡΙΣ, είναι κάτι που βοηθάει τη διοίκηση να βελτιώσει τις υποδομές, βοηθάει επίσης να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια ε, της ε, μεταφοράς μέσω εσωτερικής ναυσιπλοείας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που το κάνουν όμως αυτό. Υπάρχουν νέα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή και που αναπτύσσονται. Κάποια ευρωπαϊκά project για τη δημιουργία νέων βάσεων δεδομένων να υπάρχει ένα logbook για τα πλοία αυτά, παραδείγματο χάρη, μια σειρά ψηφιακά εργαλεία λοιπόν που θα βοηθήσουν μια πιο αποτελεσματική διαχείριση, μια πιο φτηνή επίσης ε, διαχείριση και μια πιο γρήγορη διαχείριση για όλους. Όταν μιλάμε για καινοτομία, εννοούμε και, και, ε, και πιο καθαρά πλοία. Και πρέπει βεβαίω αυτά τα πλοία να γίνουν όλο και πιο αυτόνομα. Συνεχίζονται οι εργασίες. Υπάρχουν κάποια σχέδια αυτή τη στιγμή σε πιλωτική φάση που δείχνουν ότι είναι εφικτό ε, μεσοπρόθεσμα να εφαρμοστούν. Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις για το μέλλον, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ε, τις υποδομές εσωτερικής ναυσιπλοείας και βεβαίως συνθήκες ναυσιπλοείας. είναι προβληματικές συνθήκες για την ηρεμική κυκλοφορία, την κυκλοφορία μικρών πλοίων πολλές προς μήνες του χρόνου. Έχουμε επίσης κατά νου και το πρασίνισμα του στόλου. Όταν μιλάμε για πρασίνισμα δεν σημαίνει αυτό απλά να μειωθούν οι εκπομπές του άνθρακα. Θέλουμε να μειώσουμε και τον θόρυβο, την ηχορύπανση δηλαδή. Επίσης ε, μιλάμε και για τα μελλοντικά πλοία που δεν θα είναι μόνο πιο καθαρά, αλλά θα βρεθούν περισσότερες ψηφιακές λύσεις, ε, αυτοματοποιημένες. Αυτά είχα ετοιμάσει εγώ για σήμερα, για την ε, καινοτομία στον τομέα της τεχνικής Ευχαριστώ τον κύριο Ντουράτσικ, Ντουράτσικ θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τούρι Φιωρίτο, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εσωτερικών Λιμένων. Κύριε Φιωρίτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Ρικέ. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση σήμερα. Εκπροσωπούμε πάνω από 200 λιμένες, εσωτερικούς λιμένες ε, στην Ευρώπη σας... Ε, εντάξει, με ακούτε τώρα. Θα νομίζετε ότι δεν ξέρω αυτά. Αλλά Σα είπα ότι όλου του λιμένε ε, μπορείτε να του βρείτε στι εσωτερικέ πλούτε οδού και θα σα ε, παρουσιάσω κάποια παραδείγματα για το τι κάνουμε στο διατροπικό σύστημα. Ο ρόλο μα είναι ε, να φέρουμε μαζί την εσωτερική νευσιβλοή με άλλου τρόπου μεταφορών και θέλουμε να έχουμε καλύτερε και πιο πράσινε μεταφορέ. πράσινες Το πρώτο μου παράδειγμα εδώ είναι το λιμάνι τη Λιαγής έχει ένα πολύ, ε, μια πολύ μεγάλη εγκατάσταση που τη βλέπετε εδώ. Trilogy Port λέγεται και ε, βλέπετε ότι δεν μπορούμε να εξετάζουμε μόνο τη δική μας περιοχή, ότι πρέπει να βλέπουμε όλο το δίκτυο εδώ. Βλέπετε ότι όλη μέρα της επικεντρώνεται στο να έχει σημεία πρόσβαση από τρία διαφορετικά λιμάνια, το Ρότερνταμ και την Δουκέρδη ε, και άλλο ένα λιμάνι. Έχουμε τρεις τρόπους μεταφοράς και επικεντρώνεται και σε τρεις διαφορετικές αγορές και τα μοδοποιεί όλα αυτά και τα φέρνει σε πολλές εταιρείε και επιτρέπει στην παγίωση των περιπτωματικών μεταφορών και να έχουμε περισσότερα κέρδη αποδοτικότητας και ταυτόχρονα Υπάρχει και το αεροδρόμιο της Λέγης, που είναι το 8ο ε, μεγαλύτερο αεροδρόμιο κάργο, το πραγματικό αεροδρόμιο στην ε, Ευρώπη και ίσως ε, είναι το μόνο που έχει μία διάσταση ε, τέταρτο διατροπική. Και βλέπετε εδώ τα εμπορευματοκιβώτια, γιατί τα εμπορευματοκιβώτια είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο μεταφορών εντός των διατροπικών μεταφορών. Και βλέπουμε ότι όλα είναι και περισσότερο χρησιμοποιούνται κοντέινερ. Ένα άλλο παράδειγμα για το τι ε, κάνουμε τι κάνουν οι εσωτερικοί λιμένες είναι ότι εξετάζουμε τέσσερα ποτάμια. Καταρχήν το πρώτο παράδειγμα αριστερά βλέπετε το Ροδανό και τα σχετικά λιμάνια ε, και εργαζόμαστε εκεί για να υπάρξει συντονισμό των λιμένων με τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα δημιουργούν νέα τέρμινα, νέα τερματικά πάνω και κάτω στο ποτάμι γιατί εδώ έχουμε και δύο διαδρόμου στεντή που διασταυρώνεται και αν δούμε το Δούναβι βλέπετε ότι θα ξεκινήσει το δίκτυο λιμένων του Δούναβη. Πολύ σύντομα πολλά λιμάνια στο Δούναβη συνεργάζονται για να δουν τι μπορούν να κάνουν για να αυξήσουν ε, την ε, μετάβαση στις διατροπικές μεταφορές, γιατί η προκλήση είναι ότι υπάρχει έλλειψη σύνδεση στα λιμάνια. Δεν ε, συνδέονται όλα τα λιμάνια με το σιδηρόδρομο, λοιπόν. Και δεύτερον, αντιμετωπίζουμε και το εξή θέμα. Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ε, την δυνατότητα ναυσιπλοεία στο Δούναβι πάντοτε και αυτό είναι δύσκολο για να προσελκύσουμε ε, νέε επιχειρήσει. Όμω προσπαθούν ε, τα ε, λιμάνια να προβούν σε ένα streamlining των διατυπώσεων γιατί ο μόνος τρόπος που μπορούν να ανθίσουν τα λιμάνια είναι να συνεργάζονται. Αυτό κάνουμε σήμερα και τώρα θα σας πω τι κάνουμε σήμερα για το μέλλον. Η ψηφιοποίηση αναφέρθηκε ήδη μερικές φορές, είναι το πιο σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά ε, από αυτά που κάνουμε. Βλέπετε το Port Forward, είναι ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα που τρέχει σε πολλά λιμάνια. Θα επικεντρωθώ στο Μακτεμπούργο και εδώ συλλέγουμε στο εντός του λιμάνου όλα τα δεδομένα, τι περιλαμβάνεται στην παραδειγματοκιβώτη και επιτρέπει έναν ταχύ σχεδιασμό εντός του λιμανιού αλλά και σε διατροπικό επίπεδο το RPIS ε, ε, αποτελεί ε, ουσιαστικά ένα τμήμα των συστημάτων RIS εδώ. Ξεκινάμε από το Λουμπιντισχάφεν και φτάνουμε μέχρι τη Βασιλεία. Εδώ έχουμε καταρθώσει να συλλέξουμε όλα τα δεδομένα για τους ελιμενισμούς και τις πληροφορίες σχετικά με τα κοντέινερ και σχεδιάζουμε ποια σκάφη Πώ πρέπει να κυκλοφορήσουν τα σκάφη και για να καταπολεμήσουμε τη συμφόρηση, αλλά και να βρούμε τι καλύτερε διατροπικέ λύσει για μια συγκεκριμένη μεταφορά. Βλέπουμε ότι οι εταιρείε χρησιμοποιούν ε, τι πληροφορίε από το RPIS για να σχεδιάσουν τι δραστηριότητε του εντό του τερματικού Του ξέρει ότι το σκάφο παραδείγματο χάρη, έρχεται στο λιμάνι γιατί έχει ήδη ζητήσει την ελιμινιστή στο λιμάνι σου και μπορεί να έχει το φορτηγό έτοιμο μέσα σε ένα λεπτό. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περιμένει 30 λεπτά όπω ε, συμβαίνει μερικέ φορέ άλλα πράγματα που εξετάζουμε. γιατί όπως σας είπα τα βλέπουμε από άποψη δικτύου, είναι ε, η πρωτοβουλία της ε, ζώνης που συνδέει την Ευρώπη με την Κίνα. Ε, ένας, μια δόση, μια ζώνη και μπορούμε έτσι ε, στη συνέχεια να ομαδοποιήσουμε τα εμπορεύματα στην Ευρώπη και να τα οθήσουμε προς την Κίνα και τη Ρωσία και άλλε αγορέ στην κατεύθυνση αυτή και έχουμε νέες δυνατότητες αποδοτικότητας. Μας βοηθάμε τη βιωσιμότητα και ένα ακόμη και τώρα αυτό είναι πολύ μικρό τμήμα τη αγοράς, πιστεύουμε ότι θα μεγενθεί τα επόμενα έτη. Λιόν, το Μανχάιμ, η Λιέγη και άλλα λιμάνια συμμετέχουν εδώ. Και τώρα για το τελευταίο σημείο θα πρέπει να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη μετάβαση στις διατροπικές μεταφορές. Αλλά χρειαζόμαστε να είναι συνδεδεμένα διατροπικά τα λιμάνια μας και κατόπιν χρειαζόμαστε υποστήριξη από την εθνικέ κυβερνήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεν υπάρχει πάντοτε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε με μια πιο γενική έννοια, δηλαδή να έχουμε ένα σκεπτικό που να αφορά το δίκτυο. Αισθανόμαστε ότι οι αποφάσεις Ε, πρέπει να λαμβάνονται, με ε, έναν απλό τρόπο που λαμβάνει υπόψη μόνο το ε, ένα, ένα είδο μεταφορά, αλλά θα πρέπει να τα εξετάζουμε όλα. Επίση, χρειαζόμαστε υποστήριξη και από το εθνικό επίπεδο και να διασφαλίσουμε και τη δυνατότητα ναυσιπλοεία στο Δούναβι. Αν, μπορείς να αν δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι μπορεί να κυκλοφορήσει καθόλου το έτος, ε, δεν ε, μπορείς να δεστροποιηθείς. Επίσης για μας είναι η οδηγία για τι συνδυασμένε μεταφορέ Υποστηρίζουμε τη θέση του Κοινοβουλίου και χαίρομαι για τη δουλειά του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Όμως μας ανησυχούν οι τελευταίες εξελίξεις ε, που ακούμε από το Συμβούλιο γιατί φαίνεται να πηγαίνουν προ μια διαφορετική κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ κύριε Φιωρίτο. Και για να τελειώσουμε να δώσω το λόγο στον κύριο Σούλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Συγγνώμη που άργησα, δεν με βοήθησε η κίνηση στους δρόμους δυστυχώς. Συνδέσεις μεταξύ διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Τι, τι εννοούμε. Τι μεταφέρεται εμπορευματοκιβώτια, χίδιν φορτίο που μεταφέρεται προς τον ε, προορισμό αλλά και αναμεταφορές και τα project cargo. Ξεκινώ με τα τελευταία. Είναι το, τα, βαρέα ε, φορτία χίδιν που δεν μπορούν να μεταφερθούν οδικώς γι' αυτό και επιλέγονται άλλοι τρόποι μεταφοράς, μεταφοράς προς τον τελικό προορισμό είναι κάτι που υπάρχει αλλά πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Άλλωστε υπάρχει και η δήλωση του Υπουργού Μεταφορών μας η οποία ε, ανέφερε ότι τα βαρέα φορτία στους δρόμους, στο δικό δίκτυο το καταστρέφουν. Γι' αυτό και πρέπει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος αυτών των βαρέων ε, φορτίων να μεταφερθεί στις πλωτές οδούς. Να περάσω όμως και σε κάτι πιο θετικό, τα κοντέινερ. Βλέπουμε ότι είναι χαμηλή η στάθμη στο Ρήνο και σε, άλλους, σε άλλα ποτάμια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι η εφοδιαστική αλυσίδα αμέσως ε, αναζήτησε άλλες ε, οδούς μεταφοράς, γιατί δεν γινόταν να χρησιμοποιηθούν τα ποτάμια. Ε, χρησιμοποιήθηκαν στον, ε, σε μεγάλο βαθμό τα τερματικά εκεί όπου υπήρχε ικανή στάθμη υδάτων, όπως για παράδειγμα στη Λιέγη, μεταφέρονταν τα εμπορεύματα σε φορτηγά μέχρι το σημείο όπου μπορούσαν πάλι να φορτωθούν σε εσωτερικά πλοία. Στις ε, μεγάλες ε, οδούς λοιπόν ε, στην Ευρώπη, στις μεγάλες διαδρομές, Βόρεια Θάλασσα Άλπης, Βόρεια Θάλασσα Μεσόγειας, Ρήνος, Δούναβης, ήδη γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλά δεν είναι αρκετές. Πρέπει να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο και να συμπεριλάβουν και τους άλλους διαδρόμους μεταφορών. Κάτι που έχουμε δει επίσης στην εμπειρία μας είναι σχετικά με τις διασυνδέσεις υπήρχε το ε, σειροδρομικό ατύχημα στο Ράστατ πέρσι επρόκειτο για ένα φορτίο το οποίο επρόκειτο να μεταφερθεί με, το σιδηρόδρομο δυστυχώς όμως δεν υπήρχαν αρκετές, ε, αρκετοί πόροι δεν υπήρχε αρκετή χωρητικότητα δηλαδή για να εξυπηρετηθεί εκείνη η ανάγκη μόνο από τις ιδεοδρομικές μεταφορές χρειαζόταν περισσότερο, ε, περισσότερες εσωτερικές πλωτές οδοί δηλαδή. Τι πρέπει να γίνει, να αναπτυχθούν αυτές φυσικά. Επίσης, πρόβλημα είναι το γεγονός ότι πολλές φορές μεταφέρονται από το ένα τερματικό στο άλλο άδεια εμπορευματοκιβώτια ε, σε πολύ μικρές αποστάσεις, 20, 30, 50 χιλιόμετρα. Και εκεί είναι ε, περιπτώσεις όπου πραγματικά μπορούν να γίνουν προσπάθειες για να διασυνδεθούν καλύτερα τα τερματικά. Γιατί θα ωφεληθούν πολύ. Έχουμε λιγότερες εκπομπές στις ε, πόλεις, θα έχουμε δηλαδή λιγότερες εκπομπές, ε, θα αποσυμφορηθούν ε, τα οδικά δίκτυα. Αυτά γίνονται και θα γίνουν τα επόμενα χρόνια, αλλά πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες. Από την πλευρά της ε, ναυσιπλοείας, εγώ εκπροσωπώ τον κλάδο, το ξέρετε, ε, πρέπει να σας πω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες συζητήσεις, περισσότερη δικτύωση. Χρειάζεται να ενισχυθεί και να εντυθεί ε, η συνεργασία μεταξύ των τομέων. Η εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει πραγματικά να λαμβάνει υπόψη τις, τις πολυτροπικές ή σύγχρονα, σύγχρονες παράλληλες δηλαδή μεταφορές. Αφενός δηλαδή μπορούμε να συνεχίζουμε να ανταγωνιζόμαστε προς όφελος όλων, αλλά όταν το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες πρέπει να αξιοποιούνται όλοι οι πόροι, όλοι οι διάδρομοι. Δεν θα επαναλάβω αυτά που αναφέρθηκαν για τα έγγραφα που συνοδεύουν τα φορτία. Πάντως μεγάλο μέρος της ε, κυκλοφορίας που υπάρχει ήδη σήμερα εμποδίζεται από αυτήν την ε, ε, μονόπλευρη σκέψη. Πολλές φορές υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι αξιοποιούν ή χρησιμοποιούν μόνο το οδικό δίκτυο. Τα φορτηγά, γιατί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν και εσωτερικές πλωτές ε, οδοί ή πολυτροπικές μεταφορές. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν ε, στοχευμένα συνέδρια, συμπόσια, ώστε να, να γνωριστούμε, να μιλήσουμε ο ένας με τον άλλον ή ε, οι διάφοροι κλάδοι μεταξύ τους, ώστε να φωτίζονται οι διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν. Χρειάζεται να οργανωθούν τέτοιες προσπάθειες. Τέλος. Μιλήσαμε και για, για τα ηλεκτρονικά έγγραφα. Αυτό που θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ και θα θέλαμε να κάνουμε έκκληση γι' αυτό ε, θα ήταν να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία ε, διασύνδεσης με ηλεκτρονικές πλατφόρμες άλλων κλάδων. Αναφέρθηκαν αυτά. Αλλά αυτό που δεν έχει αναφερθεί είναι το DTLF, συνδυαστικά προγράμματα που βρίσκονται ήδη υπό, σε φάση υλοποίησης, και που αφορούν ε, την, πλοήγηση. Εγώ θα έλεγα ότι τα DTLF, το DINA, όλα αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να συνδυαστούν, να συνδεθούν μεταξύ τους, γιατί είναι κρίμα να μην αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες που παρέχονται. Πολλές φορές γίνονται εκκλήσεις για νέες υποδομές. Εμείς ε, λέμε ακριβώς αυτό, ας φτιάξουμε τις υποδομές μας προτού εμφανιστούν, ε, ε, ε, εμφανιστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης, παρατηρούμε ότι σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης στην Ευρώπη υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Εκείνοι που ασχολούνται με τι εσωτερικέ πλωτέ οδού, με την εσωτερική πλοία, ασχολούνται με αντίστοιχου συναδέλφου του. Εκείνοι που ασχολούνται με το δικό δίκτυο, ασχολούνται μόνο με, το, με εκείνου που εμπλέκονται στο δικό δίκτυο. Πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν και πολλές ε, τοπικές αρχές. Πώς μπορούν να συνδυαστούν, τι μπορεί εκτός από τους δρόμους, από τους αυτοκινητοδρόμους, πώς μπορούν και τα ποτάμια, οι εσωτερικές πλωτές οδοί να αξιοποιηθούν για να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία και να περάσουμε σε αυτό το επόμενο στάδιο των μεταφορών. Euh, Ευχαριστώ τον κύριο Σούλτς και τώρα θα ακούσουμε τα σχόλια και τις ε, παρατηρήσεις των βουλευτών. Ο κύριος Βιμ Παντενκάμπ πρώτα. Δύο-τρία λεπτά παρακαλώ, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρικέ. Λοιπόν, είναι πολύ Ολλανδόφωνοι εδώ σήμερα, οπότε θα μιλήσω τη μετρική μου γλώσσα. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να επανέλθω σε αυτό το πέρασμα από το ε, έναν τρόπο μεταφοράς σε άλλο και στον πολυτροπικό τρόπο μεταφορών τέλο πάντων ε, βλέπουμε όμως ότι τελικά αυτά δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά και αντίθετα από τα που λένε οι φίλοι μας οι πράσινοι ε, θα πρέπει νομίζω αυτό το στόχο να τον θέσουμε και να επιμείνουμε αυτό το πέρασμα στο πολυτροπικό, στις πολυτροπικές μεταφορές να, να γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για αυτές τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Έχουμε πλέον μια κάποια εμπειρία στον τομέα των εσωτερικών ε, της εσωτερικής ναυσιπολογίας ε, και ξέρουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για πολυτροπικό πολυτροπικές μεταφορές έγινε αναφορά στα interface προηγουμένως κυρία Σκέπεν επίσης αναφέρθηκε στην COP21 διότι και εκεί υπάρχει ένα περιβαλλοντικό ζήτημα το οποίο έτσι κρέμεται πάνω από το κεφάλαιο κεφάλια μας έτσι με σχετικό τρόπο καλό είναι ε, ότι αναφέρθηκαν όλα αυτά. Υπάρχει και το ψήφισμα του Φεβρουαρίου. Όλα πήγαν καλά, αλλά όπως ξέρετε καλά τα ψηφίσματα, όμως θα πρέπει να δούμε πώς συγκεκριμένα τα επόμενα πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχοληθεί με την ε, εφαρμογή ε, του ψηφίσματος αυτού. διότι ότι στα λόγια είμαστε καλοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καινοτομία, Συχνά στον κλάδο μας λένε για πλοία ε, που είναι 20 έως 30 ετών, ε, πλοία που δεν είναι πολύ ε, έτσι, παλιά, αλλά χρήζουν εξχρονισμού, ανανέωσης και αυτό έχει κόστος. Πώς σκοπεύετε να το ενεργοποιήσετε αυτό. Ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η σύγχρονη ναυσιπλοεία απαιτεί χρήση, σύγχρονο εξοπλισμό, ηλεκτρονικό μεταξύ άλλων, Πώς λοιπόν σκοπεύετε να το κάνετε αυτό σε μια μεταβατική φάση και πώς σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε αυτές τις ε, ε επενδύσεις. Μπορούν βεβαίως να γίνουν κάποιες ε, τροποποιήσεις και μετατροπές, αλλά οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλες για να αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Έχουμε εδώ έναν εκπρόσωπο από την Πολωνία στο φόρουμ αυτό. Διαπιστώνω όμως ότι και στις κάτω χώρες όλο και πιο συχνά έχουμε Πολωνούς εργαζόμενους. Ε, οι Ολλανδοί είναι όλο και πιο επιφυλακτικοί να εργαστούν ε, σε αυτά τα πλοία. Και φτάνω το τελευταίο σημείο. Ε, το θέμα της φήμης του κλάδου αυτού, της εικόνας του, είναι κάπως εύθραστη αυτή η εικόνα. Υπάρχουν πολλές οργανώσεις που εκπροσωπούν την εσωτερική ναυσιπλοεία και αν το συγκρίνουμε αυτό με άλλους τομείς, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Αυτή λοιπόν η εικόνα θα πρέπει να επανεξεταστεί, θα πρέπει να βελτιωθεί. Χρειάζονται βέβαια προσωπικότητες όπως ο κύριος Φιωρίτο προφανώς, όμως δεν φτάνει ο κύριος Φιωρίτο. Δυστυχώς αυτός ο κλάδος ε, είναι, δεν είναι πολύ γνωστός, ε, δεν είναι στην επικαιρότητα, πρέπει να του δοθεί έτσι μια πιο ελκυστική εικόνα και απευθύνομαι βέβαια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση προηγουμένω. Πρέπει να προχωρήσουμε. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η ψηφιοποίηση θα αφορά το σύνολο των οδικών μεταφορών. Ε, έχει γίνει αναφορά στο διοικητικό ε, σκέλος και τα ωφέλη μιας ηλεκτρονικής ε, διαχείρισης. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε και αυτό, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι η φήμη, είναι η εικόνα του κλάδου αυτού. Ο επόμενος ομιλητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα... Και εγώ, θα ήθελα και εγώ να μιλήσω Ολλανδικά, όπως ο συνάδελφος. Ένα ερώτημα ε, διτό. Πρώτα απ' όλα, αυτή η ακρόαση είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτός ο τύπος μεταφορών έχει τεράστιες δυνατότητες ε, και σε επίπεδο ασφάλειας, βιωσιμότητας, αποτελεσματικότητας και αυτά είναι σημαντικά ατού τα οποία θα πρέπει να τα βάλουμε μπροστά. Ε, ιδιαίτερα εφόσον λάβουμε υπόψη μας και την ε, αυτόνομη, τις αυτόνομες μεταφορές έγινε αναφορά στην κλιματική αλλαγή και στην καταπολέμησή της, στα σχετικά προβλήματα. Είναι αλήθεια ότι η ξηρασία πέρυσι το καλοκαίρι αλλά και άλλα φυσικά φαινόμενα τα οποία ε, ζήσαμε, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες. Αλλού είχαμε πολύ χαμηλό επίπεδο υδάτων. Όλα αυτά δημιουργούν, είναι πραγματικές απειλές για αυτή τη μορφή μεταφορών. Ε, θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας και θα ήθελα να ζητήσω από τους εμπειρογνώμενους που είναι εδώ σήμερα να μας πούν ποια είναι η δική τους προοπτική για το μέλλον. Πώς δηλαδή συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσουμε τις συγκεκριμένες προκλήσεις στο συγκεκριμένο κλάδο. Ε, είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Και ένα δεύτερο ερώτημα τώρα Υπάρχουν μια σειρά από κενά τα οποία είναι γνωστά από όλους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα μπορεί να συνεισφέρει να καλυφθούν τα κενά αυτά. Μιλάμε όλο και πιο συχνά για ψηφιοποίηση, μιλάμε για την σημασία της βιώσιμης αποτελεσματικής διαχείρισης των πόλεων. Ίσως λοιπόν μέσω αυτού του πολυτροπικού ε, τρόπου μεταφορών θα μπορούσαμε να δούμε και τι γίνεται με τι υποδομέ και τις ανάγκες σε οι οποίες εξελίσσονται. Ε, διαπιστώνουμε παραδείγματο χάρη στη Φλάνδρα ότι αυξάνεται η μεταφορά μέσω παλετών. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει και ε, να αλλάξουν οι προδιαγραφές των, των χώρων αποθήκευση. Ε, θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε και αυτό κατά νου τι μπορεί να γίνει τα επόμενα 5-10 χρόνια ε, σε αυτόν τον τρόπο μεταφοράς και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό και σε επίπεδο αποθήκευσης. Αυτό θα μας βοηθήσει να ε, είμαστε και πιο στοχευμένοι στις επενδύσεις μας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα γιατί πρέπει να πάω σε φορές άλλη επιτροπή. Τρία ερωτήματα. Πρώτον, επειδή πέφτει η στάθμη των υδάτων στα ποτάμια, πόσο μπορεί να πέσει χωρίς να εμποδιστεί ουσιοδός ε, η δυνατότητα μεταφορών εμπορευμάτων. Υπάρχει κάποιο, κάποιο όριο κάτω από το οποίο δεν μπορούν να γίνουν μεταφορές. Δεύτερο ερώτημα. Γίνονται αρκετά για να διαμορφωθούν υποδομές με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανασηκωθούν ε, οι γέφυρες που υπάρχουν για να μπορούν για παράδειγμα να μεταφερθούν και τρει σειρέ ε, ε, εμπορευματοκιβωτίων. Τρίτο ερώτημα. Ηλεκτρι... ηλεκτρονικέ επικοινωνίες. Έχουν όλα τα σκάφη, τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά και μεταξύ τους και με τις λιμενικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ κύριο Κράμερ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές μας για τις ε, παρουσιάσεις τους. Ε, ο, ο κύριος Βάντεκαμπ ρώτησε τι λένε οι πράσινοι για τις ιστορικές πλωτές οδούς. Εμείς είμαστε υπέρ, υπό δύο προποθέσει να μειωθούν ε, οι εκπομπές και να προσαρμοστούν τα πλοία στα ποδάμια και όχι το αντίθετο. Πρέπει να διδαχθούμε και από το παρελθόν. Εγώ πριν από 25, 35 χρόνια πήγα από το Ingolstadt στη Μαύρη Θάλασσα και κάθε τόσο, κάθε 5 λεπτά έπρεπε να... Ε, ε, μετακινείται το, το πλοίο προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει ε, τις, ε, τα κύματα. Ενώ πριν από λίγο καιρό ήμουνα στον, ε, στο Δούναβι ε, και είδα τρία τεράστια πλοία να κυκλοφορούν. Τι θέλω να πω, υπάρχουν αρκετές υποδομές αλλά δεν αξιοποιούνται στο έπακρο. Στην ε, Γερμανία ε, λεγόταν για καιρό ότι όταν θα συνδεθεί ο Δούναβη με το Ρήνο θα λυθούν όλα μα τα προβλήματα. Και μετά ήρθε ο Υπουργό Μεταφορών που είπε ότι ήταν η μεγαλύτερη ανοησία το σχέδιο αυτό, το πρόγραμμα αυτό που είχε εξαγγελθεί. Γιατί, διότι έγιναν επενδύσεις ε, στις υποδομές, καλό για τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά η εσωτερική ναυσιπλοεία δεν ωφελήθηκε καθόλου. Και ε, να σας πω, ο μόνος πραγματικά βιώσιμος τρόπος μεταφορών είναι η ποδηλατόδρομη. Και εγώ την έχω κάνει αυτή τη διαδρομή και δεν χρειαζόταν εσωτερική ναυσιπλοεία. Επίσης μετά την ενοποίηση της Γερμανίας ε, υπήρχε ένα, το πρόγραμμα 17, το έργο 17, το οποίο προέβλεπε ότι θα συνδεόταν με ποτάμι εσωτερικό ε, το Βερολίνο με το Ανόβερο. Εγώ τότε είχα πει ότι πρόκειται για άλλη μια τέτοια ανοησία, όπως η περισυνδεση σύνδεσης Δούνα Βυρίνου. Αλλά χρειάστηκαν πάλι 15-20 χρόνια μέχρι να εγκαταλειφθούν αυτές οι ανοησίες δεν χρειάζεται να περνάνε τόσο πολλά χρόνια. Μπορούμε να, να διδασκόμαστε και από τα λάθη μας και από τις εμπειρίες μας. Πώς θα κάνουμε πιο ελκυστική την εσωτερική ναυσιπλοεία. Είπατε κι εσείς κάποια παραδείγματα. Υπάρχει για παράδειγμα ήδη διαδρομή μηδενικών εκπομπών. Γιατί χτίσανε μέχρι και ανεμογεννήτριες ε, οι οποίες τροφοδοτούν τα σκάφη και έτσι μηδενίζονται οι εκπομπές ή επίσης η ψηφιοποίηση που είναι πάρα πολύ σημαντική αλλά να μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη το 80% των εμπαρευματικών μεταφορών ε, που πραγματοποιούνται γίνονται στο Ρήνο. Είναι μεγάλος, βαθύς ε, ποταμός, πλατής ποταμός και φυσικά συνδέεται και με τον ωκεανό. Αυτό ναι, αλλά τα διάφορα έργα διαπλάτησης του Έλβα ή του ποταμού Όντερ. Όλα αυτά δεν έχουν ε, αξία στην πραγματικότητα γιατί μιλάμε για μείωση στην ουσία των εμπαρβηματικών μεταφορών. Εγώ μπορώ να σας πω ότι θέλω να σας κάνω έκκληση. Μην λέτε ότι χρειαζόμαστε νέε υποδομέ, οι οποίε θα μα λύσουν ω πανάκια όλα μα τα προβλήματα. Δεν συμβαίνουν έτσι. Πολλέ φορέ δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα, γιατί μπορεί απλώ να εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο τα λόμπι του, του κατασκευαστικού κλάδου. Φυσικά, πολυτροπικέ μεταφορέ, βιωσιμότητα, αλλά και εδώ είναι το σημαντικό, χρειαζόμαστε και θεμητό ανταγωνισμό. Όταν οι μεταφορέ είναι φθηνέ, ε, οι οδικέ και ακριβές οι πρέπει βεβαίω να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να αναπτυχθεί και ο σιδηρόδρομο. Και όχι μόνο ο σιδηροδρόμος και οι εσωτερικέ πλωτέ όδη. Πρέπει βεβαίω όλοι οι τρόποι μεταφορών να έχουν ίσε ευκαιρίε. Ο κύριο Λοτόφσκι για δύο-τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Άκουσα τι είπε ο κύριος ε, Ντεκάντε. Όμως δεν θα ήθελα, να πω ότι ε, δεν έρχονται οι εργαζόμενοι από την Πολωνία στο Βέλγιο ε, γιατί ε, τεμπελιάζουν στη χώρα τους. Απλώς στην Πολωνία εδώ και πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 70, έχουμε εγκαταλείψει τη, αυτόν τον τρόπο μεταφορών. Όμως οι σχολές παρέμειναν. Έχουμε πολύ καλές σχολές εσωτερικής νευσιπλογίας και στη δική μου εκλογική επικράτεια. Όλοι έχουν διπλώματα, αποφυτούν από τις σχολές, αλλά δεν μπορούν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα στην Πολωνία γιατί είναι εγκαταλελειμμένες οι υποδομές και γιατί εγκαταλείψαμε αυτό το είδος μεταφορών. Αλλά εδώ και τέσσερα χρόνια η πολωνική κυβέρνηση πάλι έχει εστιάσει στην ανάπτυξη ε, αυτού του είδους μεταφοράς της εσωτερικής ναυσιπλοείας ε, και έχουμε ε, και ένα πολύ μεγάλο ποταμό στην Πολωνία ο οποίος είναι πλωτός σε πολλά σημεία του, αλλά δεν χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις για να καταστεί πλωτός όλος ο ποταμός. Υπάρχει και το κανάλι του Μπέντικος που ε, συνδέει τον Όντερ με τον Βιστήλ και η γεωγραφική θέση του Μπέντικος θα μας επέτρεπε σε αυτή την περιοχή να κατασκευάσουμε ένα πολυτροπικό λιμάνι που θα μπορούσε να αποτελεί σημείο εισόδου για τα διάφορα λιμάνια της Βαλτικής. Και θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεται για την προοπτική αυτή ο κύριος Ντούρατσικ. Θα έπρεπε να υποστηρίξουμε μια τέτοια ιδέα. από τη στιγμή που μιλάμε για τα δίκτυα TNT. Και έχω και μια ερώτηση και για τον κύριο Φιωρίτο. Πολύ σύντομα θα έχουμε μια αναθεώρηση των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και πριν λίγο ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχιστεί το πρόγραμμα αναείδες Εσείς ε, τι περιμένετε από τη δική μας Επιτροπή Μεταφορών, τι περιμένετε από το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις επενδύσεις σε νέες υποδομές. Ξέρω ότι αυτές οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνουν μέσω των Ευρωπαϊκών ταμπίων, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και εθνικά κονδύλια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Σλοτόσκι. Δεν θα πάρω εγώ το λόγο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, όμως θέλω να αναφερθώ σε δύο θέματα. Στο θέμα της ε, δυνατότητας πλευσιπλοείας ε, αν υπάρχουν λύσεις και γιατί φαίνεται να επιδεινώνεται το πρόβλημα και ένα άλλο θέμα που δεν το αναφέρουμε και πολύ συχνά, δύσκολα το συζητάμε, τα οικονομικά πλεονεκτήματα ε, αυτών ε, των μεταφορών, των ποτάμιων μεταφορών, γιατί όλοι αναφέρονται στα ωφέλη τα περιβαλλοντικά, τα ωφέλη ε, που αφορούν τις υποδομές. Αυτό είναι υποσυζήτηση, όμως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για οικονομικά ωφέλη. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μας δώσετε την αποψή σας για το θέμα αυτό. Θα ξαναδώσω το λόγο λοιπόν στους εμπειρογνώμονες. Σας ευχαριστώ που θα τηρήσετε το χρόνο, δύο-τρία λεπτά. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Η κυρία Ντεσέπερ καταρχήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της δυνατότητας ναυσιπλοείας, γιατί ασχολούμαστε με τις υποδομές σαν και κλιματική αλλαγή. Ακούγεται κάτι πολύ δραματικό, δεν είμαστε τόσο απεσιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να εργαστούμε σε δύο πράγματα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά ε, το θέμα των πληροφοριών ε, που, έχουμε από, που έχουμε από τις αρχές, θέλουμε να έχουμε καλύτερη πρόβλεψη και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και συστήματα που να μπορούμε να ανταλλάξουμε όχι μόνο με τους πλειοκτήτες, αλλά με ολόκληρο το σύστημα της επιμηλητίας και δεύτερον αυτό που αναέφερα να δημιουργήσουμε καταλύσεις υποδομές ε, για το μέλλον. Εδώ πάμε για μια αλλαγή παραδείγματο και νομίζω ότι ε, το ξέρει αυτό και ο κύριος Κάμες ε, στο ΣΕΦ, στο Μηχανισμό Συνδέεται στην Ευρώπη, θέλουμε να έχουμε αναβάθμιση της με μεγαλύτερους δρόμους κτλ. Αλλά στους μια μεταφορές, της πλωτές οδούς, ε, έχουμε κάποια συμφόρηση και έχουμε θέματα χωρητικότητα Ξεκάθαρα, επίσης, έχουμε πολλές συμφορήσεις όπου έχουμε ε, και προβλήματα με τις επιδόσεις. Τώρα, το ζήτημα ε, που έχουμε είναι ότι δεν ε, επιλέγονται αυτά τα προγράμματα απαραίτητα για συγχρηματοδότηση, γιατί συζητούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μιλάμε για συντήρηση, όχι στην περίπτωση αυτή για μας, ε, το να καταστεί κατάλληλη η υποδομή για το μέλλον και αξιόπιστη, γιατί θέλει κάποιο αξιόπιστες υποδομές 24 ώρες το 24ωρο, δεν σημαίνει συντήρηση εξετάζουμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ομαλή ναυσιπλοεία και να καταπολεμήσουμε τις ε, συμφορήσεις. Επίσης ότι προστατεύονται τα ύδατα, η βιοπικιλότητα και με την παραγωγή ενέργειας, γιατί ξέρετε έχουμε και παραγωγή ενέργειας σε κάποιους ποταμούς. Έτσι λοιπόν ε, εργαζόμαστε ε, και για το θέμα της εγκατάστασης, αλλά όλα αυτά δεν είναι απαραίτητος επιλέξιμα. Έτσι λοιπόν θέλουμε να μας υποστηρίξετε για να είμαστε σίγουροι ότι ε, το θέμα της ανακαίνησης θα είναι επίσης επιλέξιμο και δεν μιλάμε απλώς για αναβάθμιση της χωρητικότητας. Επίσης, για το θέμα των αναγκών υποδομής. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω. Βλέπουμε βέβαια ότι προσπαθούμε να πετύχουμε μηδενικές εκπομπές, αλλά βλέπουμε ότι σε μικρότερες πλωτές οδούς έχουμε κάποια νέα ενδιαφέροντα προγράμματα και έχουμε και νέα κάργο. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε μεγάλα πλοία και μεγάλες μεταφορές, αλλά βλέπουμε και μικρότερα πλοία με μικρότερα φορτία και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το μικρό το δίκτυο θα είναι αξιόπιστο μαζί με το μεγάλο δίκτυο. Και Πάλι φτάνουμε στο θέμα της αναβάθμισης ε, της ε, επίδοσης αλλά και στο θέμα του ιδιασμού. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να έχουμε αυτή τη μεταβόρτωση στις πόλεις και θα έχουμε τις συνδέσεις όταν υπάρχει ε, ένα τερματικό εκεί και ένα τερματικό αλλού έτσι ώστε να μπορούν να συνεργάζονται αυτά αλλά μιλάμε και για πολυτομεακή διάσταση. το χάρη όταν παράγεις νέα ενέργεια στους εσωτερικούς λιμένες να να την αποθηκεύσεις εκεί, αλλά να δημιουργείς και σταθμούς καθαρής ενέργειας. Ε, έτσι, ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις ε, τις διάφορες προκλήσεις. Ο κυριος Κύριος Ντούρετσεκ, δύο-τρία λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Απαντήσω πολωνικά για να είμαι πιο ακριβής. Πολλά θέματα αναφέρθηκαν. Καταρχήν, να υπογραμμίσω ότι οι ποταμοί δεν λειτουργούν μόνο ως οδοί μεταφορών, αλλά έχουν και άλλες λειτουργίες, συνδέονται και με την οικονομία, έχουν λειτουργίες που αφορούν την προστασία κατά των πλημμυρών, κατά της ξηρασίας κτλ. Όταν μιλάμε λοιπόν για ποτάμιες υποδομές, δεν μιλάμε μόνο για τις μεταφορές, αλλά και για άλλες λειτουργίες που μπορεί να έχει ένα ποτάμι και κατόπιν είναι πολύ σημαντικές ε, αυτές οι επενδύσεις. Έτσι λοιπόν οι μεταφορές όντως αλλάζουν ε, και χρειάζεται και προσαρμογή. Και το είπατε, δεν έχουμε πάρα πολλούς Πολωνούς να εργάζονται στον κλάδο. Μιλάμε τώρα εδώ για ε, αυτοματοποιημένα ή μη αυτοματοποιημένα πλοία. Και κατόπιν ε, στην Ευρώπη αυτές οι μεταφορές γίνονται όλο ένα πιο διεθνείς. Έτσι λοιπόν χρειάζονται και γλωσσικές δεξιότητες, αλλά και όχι μόνο. Και όταν μιλάμε για τις υποδομές στις πλωτές οδούς, ναι, δυστυχώς υπάρχουν σημεία συμφόρησης στην Πολωνία, γιατί διαφέρουν τα πολωνικά ποτάμια από τα ποτάμια της δύση, και αυτό δείχνει ότι αν δεν επενδύουμε το ελάχιστο στις υποδομές, δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι οδοί. Το παράδειγμα της Πολωνίας είναι ενός λιμανιού που μπλοκάρει όλη την ευσυπλοεία σε ένα ποτάμι γιατί δεν υπάρχει αρκετός χώρος και για να απαντήσω στους βουλευτές ότι αφορά στην ε, ε, ανάπτυξη ε, στο όντερ. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται μια τέτοια ανάπτυξη της ναυσιπλοείας αυτής για να αναπτυχθεί και η χώρα. Έχουμε σήμερα τις ε, μεταφορές βαρέων φορτίων που δεν μπορούν να ε, μεταφορθούν με άλλους ε, τρόπους μεταφοράς με σιδηρόδρομο ή με οδικές μεταφορές, παραδείγματος χάρη. Γιατί είναι κορεσμένοι ήδη αυτή οι τομείς. Και αν μεταφέρετε εμπορεύματα, παραδείγματος χάρη στο Γκτάνσκ, ε, θα δείτε ότι ο ποταμός ο δικός μας στην Πολωνία θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Όμως, το πρόβλημα είναι πώς βγαίνουν τα εμπορεύματα από τα τρία λιμάνια. Έτσι λοιπόν γίνονται επενδύσεις ε, πέρα του Γκτάνσκ. Έτσι λοιπόν οι διαδρομικές μεταφορές διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Σας ευχαριστώ που σεβαστικό του χρόνου, κύριος Φιωρίτο. Ευχαριστώ. Να απαντήσω κι εγώ σε κάποιες από τις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Πρώτον, για την κλιματική αλλαγή. Φυσικά μας ενδιαφέρει ο μετριασμός των επιπτώσεων, αλλά μας ενδιαφέρει και η προσαρμογή. Γιατί αν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο των Παρισίων για 1,5 βαθμό, χρειάζεται κάποιε αλλαγέ να γίνουν στον κλάδο μα και πρέπει φυσικά να προσαρμοστούμε στην ανάγκη αυτή. Και ε, υπάρχουν, για παράδειγμα, υποδομέ που λείπουν και που πρέπει να χτιστούν τα επόμενα χρόνια. Ο κύριο Βαντεκάμπ ρώτησε για το πώ θα γίνει αυτή η μετάβαση σε καθαρότερη μεταφορά. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μελέτη η οποία έχει ως στόχο να καθορίσει τις κατευθύνσεις της εσωτερική ναυσιπλοεία τα επόμενα χρόνια και πώς μπορεί να χρηματοδοτηθούν αυτές οι νέες κατευθύνσεις. Το χρονοδιάγραμμα τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω ε, της έκδοσης αυτής της μελέτης, τη, ολοκλήρωσής αλλά πολύ σύντομα θα γίνει και θα σας ενημερώσουμε. Για την εικόνα μα στην ε, δημόσια κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στι κάτω χώρε έγινε η πράσινη εβδομάδα πρόσφατα ε, να κάτι που μπορούμε να κάνουμε, αλλά το κάνουμε τοπικά. Θα μπορούσε ίσως να γίνει κάτι αντίστοιχο και ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, βλέπω ότι σας ενδιαφέρει ε, και εσά αυτό, αλλά νομίζω ότι σε τελική ανάλυση στην κάθε χώρα πρέπει να, επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Για τον κύριο Κράμερ και το Δούναβι, να σας παραπέμψω σε αυτό που είπε ο κύριος Δεσμέκε ότι αυτό που χρειάζεται είναι αξιοπιστία των επιχειρήσεων. Ε, δεν μπορεί κανείς να πλοηγείται πάνω σε ποτάμια αν αυτό είναι επικίνδυνο ή δεν είναι εφικτό για όλα τα σκάφη. Γι' αυτό και χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε αυτό το, αυτό το θέμα. Έχω πάει και εγώ σε αυτή τη διαδρομή ε, μεταξύ Ανόβερου και Βερολίνου και είδα και εγώ το ποτάμι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε και ήταν πραγματικά πολύ διαφωτιστική η εμπειρία. Μετά, για τη διαναθεώρηση των διαδρόμων TNT που ρωτήθηκα. Ε, για τους ποταμούς Βίστουλα και Όντερ πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή γιατί αυτή τη στιγμή οι δύο αυτοί ποταμοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο και ιδίως με τις νέες προσπάθειες της πολωνικής κυβέρνησης ελπίζουμε να γίνει, να γίνει κάτι τέτοιο. Αν μπορείτε να μας δώσετε και περισσότερες λεπτομέρειες θα μπορούσαμε ίσως να μπούμε και εμείς ε, σε μια πιο συγκεκριμένη απάντηση στα ερωτήματά σας. Ναι, μπορώ να χρησιμοποιήσω και από τον δικό σας χρόνο γιατί είναι λίγο ο χρόνος. Όχι, όχι, όχι, κανένα πρόβλημα. Κύριε Βάντεκαμπ, για την οικοδόμηση της εικόνας. Μας λένε πολλές φορές ότι δεν φωνάζουμε αρκετά. Γιατί θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα. Αλλά ξέρετε, η μετριοφροσύνη και η μετριοπάθεια είναι ίδιων ε, των ε, ανθρώπων από εκεί από που προέρχομαι εγώ. Εμείς ε, συνεργαζόμαστε με διάφορες δορυφορικές οργανώσεις αν θέλετε, έτσι τις αποκαλούμε εμείς ε, συνεργαζόμαστε και με τα δύο αρμόδια υπουργεία ε, και με όλους τους εκπροσώπους των κλάδων που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Πώς λοιπόν ο στόλος, ο υπάρχον που έχει ηλικία 10 έως 40 ετών πώς μπορούμε να τον εξυγχρονίσουμε. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να τον εξοπλίσουμε με εναλλακτικά καύσιμα, βιοκαύσιμα. Αυτό βραχυπρόθεσμα μπορεί να γίνει, ε, χρειάζονται κάποιες, ε, κάποιες λίγες χιλιάδες ευρώ να εγκατασταθούν κάποια φίλτρα. Αυτό είναι εφικτό. Ακόμη και το ενδεχόμενο ε, η ενδεχόμενη αύξηση του κόστους μπορεί να απορροφηθεί από την αγορά. Μακροπρόθεσμα τα, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Θα μπορούσαμε να πούμε μπαταρίες για τις μικρές αποστάσεις 100-200 χιλιόμετρα αλλιώς χρειάζεται να έχουμε μεγάλου σταθμού φόρτισης κατά μήκο των, ε, των καναλιών και των ποταμών δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ε, ουδέτερο από άποψη εκπομπών αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι το υδρογόνο αυτό είναι πραγματική ευκαιρία ε, LNG, υγροποιημένο φυσικό αέριο, ίσως αυτό να είναι κάτι εφικτό για κάποια σκάφη, αλλά η επένδυση είναι πάρα, πάρα πολύ δαπανηρή, πάρα πολύ ψηλή και επίσης ούτε αυτό το καύσιμο είναι τελείως ουδέτερο από άποψη άνθρακα. Οπότε αυτά ως προς τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Κύριε Μεσμάκερ, για το τι βλέπουμε για το μέλλον. Θεωρούμε ότι θα υπάρχουν περισσότερα σκάφη εμπορευματοκιβωτίων και εδώ θέλω να πω αυτό που είπε και ο κύριος Κράμερ. Θα προσαρμόσουμε τα σκάφη μας στα ποτάμια. Και αυτό ήδη γίνεται. Ε, τα τελευταία 15 χρόνια ε, βλέπουμε όλο και μεγαλύτερα πλοία στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Όλο και πιο ισχυρά πλοία, με μεγαλύτερες επιδόσεις. Αυτό πρέπει να σταματήσει θα πρέπει τα μελλοντικά σκάφη να ναυπηγούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στι ανάγκε του, του μέλλοντο, των φορτίων, των εμπορευματικών μεταφορών. Βεβαίω και αυτό θα απαιτήσει πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί. Τι άλλο. Νέα κανάλια. Έχω μια μεγάλη δήλωση που, θέλω να κάνω. Είπατε έτοιμο για το, για το, για το μέλλον. Οι λύσεις μας θα πρέπει να είναι έτοιμες για τις λύσεις. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει από σήμερα να ξεκινήσουμε για να καταστήσουμε τις γέφυρές μας ανθεκτικές για το μέλλον. Σας ευχαριστώ και εσούς, ευχαριστώ όλους. Δεν συζητάμε αρκετά το θέμα αυτό και έτσι μένουμε όλοι έτσι με την όρεξη να πούμε περισσότερα. Πάντως εμείς εκφράσουμε το ενδιαφέρον μας για τις ε, εσωτερικές θαλάσσιες οδούς, ε, το υποστηρίζουμε. Υπάρχουν κάποιες προκλήσεις σε επίπεδο ε, της νεωτερικότητας, συγχρονισμού. Σας ευχαριστώ όλους και τους τέσσερις Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όπως γνωρίζετε, μάθαμε όλη την περασμένη εβδομάδα την ατύχημα του ε, Boeing 737 MAX 8 με του 157 νεκρούς της Ethiopian Airlines μετά το άλλο ατύχημα, δυστύχημα της 189 θύματα τον Οκτώβριο του 2018 ε, της, Ινδονησιακής εταιρείας με το ίδιο αεροπλάνο, δηλαδή το ίδιο μοντέλο. Αυτό δημιούργησε πολλά ερωτηματικά ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και είναι κάτι το οποίο απασχόλησε την επικαιρότητα, οδήγησε σε μια σειρά από μέτρα τα συγκεκριμένα αεροσκάφη δεν μπορούν πλέον να πετάξουν. Ξεκίνησε από την Ανατολή αυτή η απόφαση προς τη Δύση. Οι Αμερικανοί αντιστάθηκαν μέχρι ένα σημείο. Τελικά όμως και αυτοί αποφάσισαν να μην επιτρέψουν αυτά τα μοντέλα του, της Boeing να ε, πετάξουν. Ευχαριστώ τον Πατρική που είναι εδώ μαζί μας και διευθύντη διευθυντής της Ευρωπαϊκής ε, Εταιρείας, ε, Ευρωπαϊκής ε, εναέρεια ασφάλειας ε, ε, σιδηρόδρομος είπα εγώ α συγγνώμη συγγνώμη είναι από την προηγούμενη συζήτηση αυτό λοιπόν ε, τον ευχαριστώ τον κύριο Κι που μπόρεσε να βρει χρόνο να έρθει να μα μιλήσει ενώ έχει φορτωμένο πρόγραμμα ίσω και ακόμα πιο φορτωμένο τώρα για να μας πει την άποψή του και να απαντήσει και στα ερωτήματά μα. τα ερωτήματα που έχουν και οι απλοί πολίτες. Διότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο και στον τομέα των αερομεταφορών αλλά και στον τομέα του κλάδου, του βιομηχανικού της αεροναυπηγικής. Ξέρετε ότι όσο διατηρείται αυτή η κατάσταση οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες παγκοσμίω. Λοιπόν, θα μας μιλήσει ο Πατρίκ για το θέμα αυτό και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τα ερωτήματα των βουλευτών. Νομίζω πως είναι ε, εξαιρετικά έτσι θερμό το ζήτημα αυτό αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Επιτρέψτε μου να περάσω στα αγγλικά. It's working, yes. Εντάξει, όλα καλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν μου το επιτρέπετε, θα κάνω την παρουσίασή μου στα αγγλικά, Μία και όλοι τεχνικοί όροι είναι στα αγγλικά. Δεν ξέρω, είναι κρίμα που θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Συγγνώμη. Θα ήθελα να ξεκινήσω βεβαίως ε, εκφράζοντας τη λύπη μου για την τραγωδία της Ethiopian Airlines 57 νεκροί αυτό το δυστύχημα. Όπως ξέρετε το 2017 ήταν το πιο ασφαλές έτος ε, για την, ε, την, ε, τις μεταφορές. Το πιο ασφαλές έτος στην ιστορία της, ε, των αερομεταφορών. Δυστυχώς όμως το 2018 είχαμε 11 δυστυχήματα με πάνω από 500 νεκρούς Αυτά τα τραγικά γεγονότα μας έστειλαν πίσω ε, σε στοιχεία που δεν είχαμε ξαναζήσει το 2015 και αυτό μας θυμίζει ότι δεν μπορούμε ποτέ να επαγρυπνούμε σε συστήματα ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά το σκάφος 302 πρόκειται για το Boeing 737 MAX ε, που είχε πιστοποιηθεί από τους ε, συναδέλφους μας η, Σικάγο, η σύμβαση του Σικάγου του 14, ε, μάλλον το 1984 προβλέπει ότι πρέπει να πιστοποιούνται από το κράτο στο οποίο βρίσκονται τα αεροσκάφια αυτά. Στην περίπτωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ε, δουλειά αυτή την έχει αναλάβει η ΕΑΣΑ. Στην περίπτωση του Boeing, έχουμε ήδη πιστοποιήσει το σχετικό αεροσκάφο, οπότε αυτή η επαναπιστοποίηση ε, ουσιαστικά ακολουθεί μια παραφέρει διαδικασία και για άλλα προϊόντα όπου ε, εμεί ε, επαναπιστοποιούμε το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Γιατί σε ό,τι αφορά τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια διμερή συμφωνία από το Μάιο του 2012, 2011 και έτσι έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο η αρχή επιστοποίησης περιορισμένο σε συγκεκριμένη ε, υπόθεση συγκεκριμένη υπόθεση για του Αμερικανού ε, στα εξή καθήκοντα. Και θα σας το δείξω τώρα εφόσον μπορέσω. Oh, yes. Easy. You do it. Thank you. So, the area... Λοιπόν, οι τομής όπου μια αρχή πιστοποίηση εμπλέκεται είναι η εξή. Στην περίπτωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ τα βλέπετε, τις βλέπετε εδώ, τομείς όπου υπάρχει μια διαφορά επί της ρύθμισης, καινούρια ή μη συνηθισμένα στοιχεία όπως νέες τεχνολογίες, καινούριε ε, μέθοδοι συμμόρφωσης ή στοιχεία τα οποία δεν συμμορφώνονται ε, άμεσα, καθώς και ευαίσθητα ζητήματα που συνδέονται με ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα ε, για ένα προϊόν το οποίο έχει παρεμφερείς παραφέρει χαρακτηριστικά σχεδιασμού. Ε, σε ό,τι αφορά την ΕΑΣΑ τώρα, εμείς εξετάζουμε τις πληροφορίες και τις επιστοποιούμε, τις πληροφορίες του κατασκευαστή. Επίσης κάνουμε τεστ πτήσεων, σε μικρότερο βαθμό βέβαια, διότι δεν, όταν δεν είμαστε εμείς πρωτεύουσα αρχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για το Boeing 737 MAX, η Boeing μας υπέβαλε τα νέα στοιχεία που σχετίζονται με αυτή τη νέα γενιά αεροσκαφών. Είναι η τέταρτη γενιά 737. Η πρώτη άρχισε να, να εμφανίστηκε το 1964. Και με βάση την παρουσίαση αυτή της Boeing και τις συζητήσεις που είχαμε την FAA και την Boeing αποφασίσαμε ε, που θέλαμε και εμείς να συμμετάσχουμε και να έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ε, παρακολούθησης. Τομείς, οι τομείς στους οποίους εμείς δεν ε, παρεμβήκαμε, βασιστήκαμε αποκλειστικά στην αξιολόγηση από τους Αμερικανούς συναδέλφους. Εμείς λοιπόν κάναμε μια ανάλυση ό,τι αφορά, τώρα θα μπω λίγο σε τεχνικά ζητήματα, έτσι, αλλά πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι στην διαχείριση των λαθασμένων παραμέτρων ε, δεδομένων ε, αεροπορικής ε, μεταφοράς. Ε, πάνω από δύο χρόνια είχαμε συζητήσει με την FAA για το θέμα αυτό και το Μάρτιο του 2017 ολοκληρώθηκαν αυτές οι συζητήσεις όταν λάβαμε επιτέλους ικανοποιητικές απαντήσεις στα αιτήματά μας. Δεν εξετάσαμε τα συστήματα ελέγχου των πτήσεων διότι αυτά θεωρήθηκαν ότι δεν επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις ή ελάχιστα επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις. Τώρα και το ατύχημα 610 ε, ε, τέλο πάντων της Lion Air εξακολουθεί να είναι υπό έρευνα, υπό διερεύνηση. Όμως η προκαταρτική αξιολόγηση και τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι υπήρχαν προβλήματα έλεγχου της πτήσης που βασίζονται ε, στο ότι κάποιοι σένσορες δεν λειτουργήσαν και βεβαίως κάποια χαρακτηριστικά ε, του ΕΜΚΑΣ δεν, ε, ε μάλλον παρουσιάσαν της λειτουργίας. Ε, μιλάμε για κάποια μικρά φλαπ που βλέπετε εδώ, που βρίσκονται στο πλάι των, του αεροσκάφους και καθορίζουν ποια είναι η κίνηση που πρέπει να κάνει το αεροσκάφος ανάλογα με τη γωνία που πρέπει να πάρει, πτώση, ανάλογα με τον αέρα, με τον άνεμο. Περνάμε στην επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια. Τώρα το MCAS, το MCAS, το, είναι ένα, μια συσκευή, ειδικά για το Max, έτσι ώστε να μπορεί, να, να, μπορεί όταν στρίβει απότομα ή όταν είναι σε χαμηλή τραχύτητα το αεροσκάφος να μπορεί να κατέβει. Είναι μια διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο αεροσκάφος για να υπάρχει και μια παρεμφερής κατάρτιση των ε, πιλότων. Όταν δηλαδή το σύστημα βλέπει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, τότε το MCAS αρχίζει να, να, να βάζει σε λειτουργία αυτό το σύστημα το nose down, δηλαδή της ε, ε βουτιάς του αεροπλάνου αυτού. Μετά τα στοιχεία που έκρυψαν από τις αρχές της Ινδονησίας που είχαν σχετικές έρευνες, η Boeing ανέλαβε μια σειρά αποδράσεις Στις 6 Νοεμβρίου υπήρξε ένα χειρίδιο OMB, Operation Manual Bulletin, δίνοντας οδηγίες ε, στο πλήρωμα να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη διαδικασία όταν ε, διαπιστώνουν ότι η ταχύτητα ε, δεν είναι αξιόπιστη. Στις 11 Νοεμβρίου η Boeing ενημέρωσε όλους τους πελάτες του Max ε, σε περιφερειακό επίπεδο μέσω πολλών μηνυμάτων δόθηκαν πληροφορίες λοιπόν για το ΕΜΚΑΣ μέσω ενός συστήματος πολλαπλών μηνυμάτων αυτά τα στοιχεία λοιπόν, αυτές τις πληροφορίες στάλησαν σε όλους τους χρήστες του 737 MAX το Νοέμβριο έγιναν αυτά η FAA που είναι η, η πρωτεύουσα αρχή επιστοποίησης μία μέρα αργότερα ε, εξέδωσε μία κατεπίγουσα οδηγία την οποία βλέπετε εδώ που λέει λίγο πολύ τα ίδια αυτή η οδηγία ενεκρίθη από την ΕΑΣΑ στις 8 Νοεμβρίου με αναδρομική ισχύ από 7 Νοεμβρίου. Ο στόχος αυτής της οδηγίας είναι να, να, να γνωστοποιηθεί στο πλήρωμα ότι εάν το ΕΜΚΑΣ αρχίσει να λειτουργεί χωρίς να του ζητηθεί να λειτουργήσει πρέπει να εφαρμοστεί μια συγκεκριμένη διαδικασία που είναι η διαδικασία του Runaway Stabilizer. Παραλλήλως, αλλά αργότερα, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο η Boeing και η FAA παρουσίασαν στην ΕΑΣΑ δύο σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό που έπρεπε να επικυρώσουμε και που αναφέρονται κυρίως στο MCAS αλλά και αναφέρονται και επίσης και στο γεγονός ότι υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ δύο σένσορων AOA και υπήρξε και σχετικό αίτημα για ε, τις απαιτήσει κατάρτισης ε, ενώπιση των αλλαγών αυτών. Με βάση την ανταλλαγή πληροφοριών με την FAA και το Boeing και μετά την ανάλυση του ατυχήματο που δεν έδειξε να υπάρχουν παρεμφερή προβλήματα με τέτοιου σένσορες ή το MCAS στον επιχειρησιακό στόλο η ΕΑΣΑ θεώρησε ότι η δράση που ανέλαβε η FAA και η Boeing, δηλαδή τα διορθωτικά αυτά στοιχεία, καλύπτουν τον επίπεδο κινδύνου, το κίνδυνο για την ασφάλεια. Με βάση λοιπόν τις δράσεις της Boeing και της FAA, τις αντιδράσεις τους, περιπτώσει, και με βάση και τον αριθμό των ατυχημάτων που περιλαμβάνουν περιεμφερή τύπου ε, γεγονότα, θεωρήσαμε ότι αυτό που μας πρότεινε η Boeing αρκούσε για να καλυφθεί ο κίνδυνος για ένα τουλάχιστον μικρό χρονικό διάστημα. Να έρθω τώρα στην απόφαση που πήραμε την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή να απαγορεύσουμε την πτήση αυτών των αεροσκαφών. Πρώτα απ' όλα, το ότι είχαμε δεύτερο ατύχημα μέσα σε πέντε μήνες, αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, είναι κάτι εξαιρετικό. Αφορούσε ένα νέο αεροσκάφος που είχε αρχίσει να λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο περίπου και αυτό βεβαίως ε, κατέστησε ακόμα πιο ανησυχητικό, ανησυχητική κατάσταση. 600.000 600 μάλλον ώρες πτήσεων είχε μόλις κάνει αυτό το αεροσκάφος 600.000 ώρες πτήσεων και κάτι για το οποίο θα χρειαστούμε κάποια υποστήριξη από, Ευρωπαϊ, από τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα αργότερα, δεν μπορέσαμε να συμμετάσχουμε στην έρευνα. Είναι αμερικανικό αεροσκάφο, το, το έχουν πιστοποιήσει οι Αμερικανοί παρότι είχαμε πάνω από 40 ε, θύματα Ευρωπαίους. Αναγκαστήκαμε να βασιστούμε λοιπόν μόνο στη δημόσια ενημέρωση και στην ενημέρωση της FAA ε, που αυτή τη στιγμή ε, ασχολείται με την έρευνα. Οπότε για μας, για μια υπηρεσία σαν τη δικιά μας, είμαστε σε μια πολύ λεπτή, άβολη θέση, δεν έχουμε πρόσβαση δηλαδή στην ίδια την έρευνα. Τρίτον, οι εμπειρογνώμονές μας ανέλησαν πολύ προσεκτικά την πορεία του αεροσκάφου της ET302 e σε σχέση με την LA610, δηλαδή της Lion Airlines, υπήρχαν διαφορές αλλά και υπήρχαν και κοινά σημεία. Και τέταρτον, όταν συζητήσαμε με τις εθνικές αρχές μετά το ατύχημα της Ethiopian Airlines, όταν συζητήσαμε με τις εθνικές αρχές και τις εταιρείες που χρησιμοποιούν τη MAX και ρωτήσαμε κατά πόσο τα πληρώματα, τα πληρώματα τους ε, μπορούν, είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα μέτρα που είχε συστήσει η Boeing λάβαμε ε, καθυσυχαστικές απαντήσεις ότι βεβαίως ενημερώθηκαν όλα τα σχετικά πληρώματα αλλά ότι στην πράξη ήταν πολύ δύσκολο να ελέγξει κανείς, να κάνει μια προσωμείωση ε, σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον τέτοιων γεγονότων. Όταν δηλαδή μόλις έχει ε, σηκωθεί το αεροπλάνο ε, και εμφανιστούν τα συμπτώματα αυτά, είναι δύσκολο κανείς να το ελέγξει αυτό σε ένα καθεστώς ε, πίεσης, ε, το πώς δηλαδή ένα πλήρωμα θα αντιδρούσει στην πραγματικότητα δεν μπορεί να δημιουργηθεί δηλαδή, με τέτοια κατάσταση ε, εικονικά. Με βάση αυτά τα τέσσερα στοιχεία αποφασίσαμε ε, να εκδώσουμε μια κατεπίκουσα οδηγία σε ό,τι αφορά τα πλοία ε, τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε, σε, σε, σε ευρωπαϊκά μητρώα ε, απαγορεύοντας το να μπορέσουν αυτά τα αεροσκάφη να πετάξουν. Αυτή η απόφαση βασίστηκε στην τεχνική και επιχειρησιακή ανάλυση, δεν την υπαγόρευσε σε καμιά περίπτωση οποιαδήποτε πολιτική πίεση. Η πρώτη μα προτεραιότητα είναι να προστατεύσουμε του πολίτε μα και όχι να κάνουμε πολιτική. Αυτή είναι η τρίτη φορά στην ιστορία τη ΕΑΣΑ που απαγορεύουμε την πτήση εμπορικών αεροπλάνων. Μετά το Falcon 7X για τρει εβδομάδε το 2011 ε, και το το 2013 για τρεις μήνες ε, το Boeing επίσης. Περιμένουμε ακόμα στοιχεία από την έρευνα. Ζητήσαμε επισήμω από τι αρχέ τη Αιθιοπία να συμμετάσχουμε ω παρατηρητέ στην έρευνα αυτή και παράλληλα συνεργαζόμαστε με την Boeing και την FAA για να αξιολογήσουμε και να εφαρμόσουμε ε, βελτιωτικά μέτρα ε, για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Η μέρες μας ακούσαν τις απαντήσεις είναι η, Ρέιτσελ Τζεσλέρ μαζί μου και ο Λοβίκ Λαό ε, που ασχολείται με τα μεγάλα ε, εμπορικά αεροπλάνα. Ε, Ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Ας ακούσουμε τώρα τις ερωτήσεις των βουλευτών. Να ξεκινήσουμε με τον Βιμ Βαντεγκάπ. Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Κυριακή. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πολύ σαφή παρουσίαση. Μιλώ πραγματικά με βαριά καρδιά όταν ε, βλέπω τα πολιτικά σχόλια που πρέπει να γίνουν ε, κατόπιν του ατυχήματος. Συνεχίζονται και οι δύο έρευνες ε, και για τις Ινδονησιακές και για τις Αιθιοπικές αερογραμμές. Και νομίζω ότι ως πολιτικοί θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα εξονυχιστικοί. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτό το αεροσκάφος έχει πιστοποιηθεί από την FAA και έχει εγκριθεί από εσά Ω ασφαλέ, Όμως πολλά προβλήματα ανέκυψαν. Η ερώτησή μου αφορά τα μαύρα κουτιά. Από ό,τι καταλαβαίνω, τα μαύρα κουτιά της στήσης αυτής τα πήγαν στο Παρίσι για περαιτέρω έρευνα. Έχετε πρόσβαση σε αυτά. Συμμετέχετε στην έρευνα των μαύρων κουτιών. Και κάτι άλλο που με εντυπωσίασε ήταν ότι διάβασα στον Ολλανδικό τύπο ότι στις 6 Νοεμβρίου ε, είχαμε ε, την επιχείρηση Manual Bulletin από την Boeing, καλά. Δεν την είχαν διαβάσει οι πιλότοι γιατί ήταν πάρα πολύ τεχνική και λεπτομερής. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτό το θέμα, αυτό το εγχειρίδιο, το επιχειρησιακό εγχειρίδιο. Είναι κάτι που είχε ε, ουσιαστικά εντυπωθεί από τους πιλότους, γιατί έγιναν πολλά σχόλια στον Ολλανδικό τύπο για αυτό το θέμα. Επίσης, ε, υπάρχει και το θέμα της ε, οδηγίας περί αξιόπλου της FAA. τη γνωρίζουν αυτή την ε, οδηγία γιατί την έχουν εντυπώσει όσοι εργάζονται στον κλάδο. Επίσης, ε, ξέρουμε κάτι περισσότερο για το εγχειρίδιο, δηλαδή ότι υπάρχει και μία ε, επικαιροποίηση του λογισμικού, του software. Και θα ήθελα να δω τι έχει να πει και η Κομισιόν. Ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλής Αεροπορίας θα έπρεπε να συμμετέχει σε αυτή την έρευνα και θα πρέπει να γίνει αυτό γιατί ε, σε αυτό το αεροσκάφο ήταν και Ευρωπαίοι πολίτε. Πρέπει να προστατεύσετε τους πολίτε μα. Επομένω, βεβαίω και πρέπει να συμμετέχουμε στην έρευνα αυτή. Χρησιμοποιείται με πολύ προσεκτικό τρόπο Τη λέξεις. Μας ε, είπατε ότι ε, ζητήσατε να συμμετέχετε στην έρευνα ε, για το αεροπορικό δυστύχημα στην Αιθιοπία, όμως δεν μας έχετε πει τίποτα για το σε ποια κατάσταση, σε ποια εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην οδηγηθούμε σε εξαγωγή συμπερασμάτων ακόμη. Ευχαριστώ, Βιμ. Ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Κύπ. Παρόμοια τα ερωτήματά μου με εκείνα του κύριου Βάντεκαμπ. Πρώτον, διαπιστώνουμε το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ανησυχητικό. Μέσα σε έξι μήνες Καταστράφηκαν ολοσχερό, είπατε εσεί. Για μένα δεν, είναι, δεν πρόκειται απλά για ολοσχερή καταστροφή, αλλά για θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων. Από αυτή την άποψη είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, πάρα πολύ σοβαρό το φαινόμενο και ανησυχητικό. Γι' αυτό και πρέπει να ασκήσουμε πιέσει, ώστε στο μέλλον, και εδώ ξεκινάει και το ερώτημά μου, ποιε θα είναι οι διαδικασίε που θα ακολουθούνται. Αν, για παράδειγμα, στι ΗΠΑ εγκρίνεται μέσω τη FAA ένα αεροσκάφο, Αποδέχεται αυτή την έγκριση αυτομάτως, αν θέλετε, η ASAA ή υπάρχει μια ξεχωριστή έγκριση τύπου. Δεύτερο, πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Αν κατάλαβα καλά από τις αναφορές στον τύπο, αυτό το MCGA, ή τέλος πάντων πώς το είπατε, αυτό το σύστημα, μου φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο διατίθεται πλέον σε επιχειρήσεις αεροπορικές που δεν, ξέρω, δεν θέλω να, να, να διασπείρω και ψευδείς ειδήσει, αλλά ακούστηκε κάτι τέτοιο στο γερμανικό τύπο ότι σε κάποιες, φορέ, κάποιες φορές δόθηκαν εγκρίσεις χωρίς να χρησιμοποιούνται οι πλέον επιμελείς ε, διαδικασίες. Πολλές φορές, δηλαδή, αντί για καταστροφικό αποτέλεσμα, ε, αναφερόταν στην έγκριση την Αμερικανική ότι το, το επιτέλεσμα θα μπορούσε να είναι απλώς επικίνδυνο. Πώς γίνεται όμως η ESA, η δική μας υπηρεσία, να αποδέχεται σχεδόν αυτομάτως ε, τις εγκρίσεις που ε, δίνονται στην Αμερική. Αν κάτι τέτοιο πράγματι συμβαίνει, θεωρώ ότι είναι πολύ προβληματικό για να μην πω και σκανδαλώδες. Τρίτο ερώτημα. Πώς γίνεται να γίνεται μια πτώση αεροσκάφους, του αεροσκάφους της ε, Lion Air, να έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα στο λογισμικό και στο μεσοδιάστημα να συνεχίζεται να, επιτρέπεται, να, επιτρέπονται οι πτήσει αυτών των αεροσκαφών σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μάλιστα όχι μόνο συνέχιζαν να πετάνε αυτά τα αεροπλάνα, έγιναν και παραγγελίε και αγορές νέων τέτοιων αεροσκαφών. Εγώ ελπίζω και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου ώστε τα, ε, τα αεροσκάφη αυτά να μείνουν ε, στο έδαφος να μην ξανασηκωθούν έω ότου διαλευκανθεί πλήρω η υπόθεση. Γιατί έρχεται και το καλοκαίρι και ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα πετάξουν στι διακοπέ του, θα χρησιμοποιήσουν τα αεροπλάνα για να πάνε στου ε, τόπου προορισμού του. Άρα το ερώτημά μου είναι, ποιο ευθύνεται για το γεγονό ότι χρειάστηκε τόσο πολύ χρόνο, μετά το ατύχημα της Lion Air και γιατί χρειάστηκε να έχουμε και δεύτερο ατύχημα έως, ως, ε, ότου ληφθεί αυτή η πιο δραστική ε, πρωτοβουλία να ε, ακινητοποιηθούν όλα αυτά τα αεροσκάφη. Δεν είναι δυνατόν δε να είναι η, η Αιθιοπία, η Ινδονησία και άλλες χώρες εκείνες οι οποίες πρώτες πήραν αυτή την ε, πρωτοβουλία. Επίσης, πώς θα, δια, θα διασφαλίσουμε, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι πράγματι με μια απλή αναβάθμιση του λογισμικού τα αεροσκάφη αυτά θα ξανακαταστούν ασφαλή. Και όπως είπε και ο κύριος Φάντεκαμπ, γιατί δεν συμμετέχει στην όλη διαδικασία η ΕΑΣΑ, τι έχει διδαχθεί, ποια είναι τα διδάγματα που έχει αντλήσει από αυτή την υπόθεση η ΕΑΣΑ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Να μην ξεχνάμε, όσο δυνηρή και αν είναι ε, η υπόθεση αυτή ότι 25.000 άνθρωποι ε, το χρόνο πεθαίνουν στους δρόμους της Ευρώπης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Στο 92% των περιπτώσεων ήταν, ε, πρόκειται για ανθρώπινο σφάλμα. Μήπως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις αερομεταφορές. Μήπως ε, απλώς ε, τα αεροσκάφη αυτά όπως έχουμε δει και σε στρατιωτικά τυχήματα τα τελευταία χρόνια πέφτουν γιατί η τεχνολογία δεν είναι επαρκής. Σα ευχαριστώ που ήρθατε εδώ κύριε και σήμερα. Δεν θέλω ούτε εγώ να εξάγω συμπεράσματα προώρα, από ό,τι φαίνεται να μπορεί να είναι αυτό ένα πολιτικό σκάνδαλο παρόμοιο με το Dieselgate και ξέρουμε έχουμε περίπου 470 μαξ ε, που λειτουργούσαν μέχρι την ακινητοποίηση και ίσως ε, πρέπει να σκεφτούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γιατί αν άρεται την εντολή αυτή τότε θα μπορέσουν να ξαναπετάξουν αυτά τα αεροσκάφη στον ευρωπαϊκό ενέργειο χώρο και θέλω να επενθυμίσω ότι πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες ε, όπως είπε και ο συνάδελφος Ισμαήλ χρησιμοποιούν ε, τακτικά αυτά τα αεροσκάφη, ε, η ε, Norwegian Airways, στην Ιταλία, άλλη εταιρεία, η Ryanair, έχει μόλις παραγγείλει 135 τέτοια αεροσκάφη και με δυνατότητα να παραγγείλει περισσότερα. Αυτό λοιπόν που κάνουμε τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι θα πρέπει ίσως να γνωρίσουμε ότι το σύστημα MCS που εξηγήσατε πάρα πολύ καλά που έχει αναπτυχθεί για εξοικονόμηση πόρων και τελικά ε, δεν θα έπρεπε να γίνει να έχει σχεδιαστεί εκ νέου αυτό το αεροσκάφο. Είναι σαφέ από τι έρευνε που συνεχίζονται ότι δεν θα έπρεπε να έχουν προσπαθήσει να επικαιροποιήσουν ε, ε, το αεροσκάφο και αν υπάρχουν νομικά ζητήματα τότε τι κάνουμε με αεροπλάνα τα οποία είχαν ένα αρχικό συνδυασμό που επικαιροποιήθηκε και έγινε αυτό για λόγους εξοικονόμηση χρημάτων. Συγγνώμη που τα λέω αυτά και έχω αυτό το πολιτικό επιχείρημα, αλλά αισθάνομαι ότι αυτό έγινε σε αυτή την περίπτωση. Αναφερθήκατε σε διάφορες ε, θέματα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, υπήρχαν ε, και κάποιες αναφορές πιλότων για το πρόβλημα, συγκεκριμένα για αεροσκάφη που δεν ε, έχουν συντριβεί ίσως Αμερικανοί πιλότοι. Όμως εσείς είχατε κάποιες αναφορές από Ευρωπαίους πιλότους ή από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων σας, γιατί είναι σαφές ότι αυτό το πρόβλημα αρχίζει να αναδύεται και πριν από το Οκτώβριο, Οκτώβριο πέρσι και σίγουρα από τότε. Και ε, μια άλλη αναφορά στο τύπο λέει ότι ε, βγαίνουν σε διάφορα μοντέλα αυτά τα αεροσκάφη και ότι εν μέρει είναι οικονομικό το θέμα. Όμως ε, οι εταιρείε μπορούν να παραγγείλουν αυτά τα αεροσκάφη με μια πιο προηγούμενη προηγμένη έννοια της ε, ε, γωνίας επίθεσης ε, για να μετριαστεί το πρόβλημα. Το γνωρίζετε αυτό το θέμα και μπορείτε να μου πείτε ποιες ευρωπαϊκές εταιρείε ή θα παρακολουθήσετε ποιες ευρωπαϊκές εταιρείες αερομεταφορών έχουν παραγγείλει τα πιο ακριβά αεροσκάφη με, με τους καλύτερους αυτούς αισθητήρε, Anglo Fatak. Επίσης, Πολύ χρήσιμα μας είπατε ότι το πρόβλημα ε, που έχετε με τις διεθνείς συμφωνίες και πώς αυτό σας δένει τα χέρια ε, και ε, συζητάτε σε επίπεδο διεθνούς δικαίου για τον αντίκτυπο, γιατί μου φαίνεται ότι υπάρχουν πραγματικά θέματα για το αν η Αμερικανική κυβέρνηση FAA έχει πλήρως συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Μπάσα, γιατί από ό,τι φαίνεται από την ανάλυση κινδύνου αφέθηκαν κάποια επίπεδα χειρισμού στην Boeing, ενώ δεν θα έπρεπε να έχει γίνει, γιατί αυτό ήταν κρίσιμο ζήτημα. Και πολύ συχνά είναι δεμένα τα χέρια σα και δεν μπορείτε να κάνετε πολλά, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα διεθνού δικαίου αυτό. Και τέλο, ε, από τον νέο βασικό κανονισμό για την ΕΑΣΑ, δυνάμει του άρθρου 1-2K έχετε το καθήκον να υποστηρίζετε ε, την ε, επιβατικό σκέλος ε, στην, ε, ε μη στρατιωτική αεροπλοεία. Και θέλω να πρακτικά να μου πείτε τι κάνετε. Ναι, προβήκατε ε, σε αυτή τη κινητοποίηση, όμω. Ε, Πολλέ φορέ ε, μπορεί να χρειάζεται να ανακλείσετε πιστοποιητικά. Και τι άλλο κάνετε για να σεβαστείτε τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 1 του βασικού κανονισμού. Ευχαριστώ, Λουσίου κύριο Κράμερ. Ευχαριστώ και για την παρουσίασή σας. Στο γερμανικό τύπο, στο Spiegel, εμφανίστηκε μια συγκεκριμένη αναφορά και εκεί αποδίδεται ε, η ευθύνη στην Airbus για τα ατυχήματα αυτά. Γιατί η Airbus, λέει, ανέπτυξε το 2010 ένα νέο μοντέλο, ε, εγκατέλειψε τις ε, ε, ε, έβγαλε λοιπόν στην, ε, στην αγορά ένα νέο αεροσκάφος. Η Boeing λόγω ανταγωνισμού επιτάχυνε τις διαδικασίες της και μέσω των αλλαγών που χρειάστηκε να κάνει για λόγους ανταγωνισμού όπως είπα δεν ενημερώθηκαν οι πιλότοι, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα, τα στοιχεία στο εγχειρίδιο και ξαφνικά η κλίση των αεροσκαφών ήταν τόσο απότομη που έπεφταν. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι η Airbus είναι καλύτερα, κάτι που η Boeing δεν μπορεί να αποδεχθεί. Επίσης, αναφέρθηκε η πληροφορία ότι πολλοί πιλότοι έχουν εκ των προστέρων ε, διαμαρτυρηθεί ότι πολλές φορές γίνονται πράγματα στα αεροσκάφη, στα πιλωτήρια, χωρίς να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Εσείς έχετε λάβει τις καταγγελίες και τι έχετε κάνει. Τέλος, Οι ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ ήταν πάντοτε πάρα πολύ αυστηρές έως το 2005. Όποτε υπήρχε κάποια αλλαγή γίνονταν πάρα πολύ ε, ενδελεχείς έλεγχοι. Μετά άλλαξαν οι κανόνες και ανατέθηκε στην ίδια την Boeing να κρίνει αν, κάτι πρέπει να, αν, κάτι, αν κάποια αλλαγή είναι ουσιώδης ή όχι. Αυτές οι αλλαγές, αυτή η χαλάρωση των κανόνων έγινε για να βοηθηθεί στον ανταγωνιστή με την Airbus η Boeing. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Θα πρέπει κάθε αλλαγή να εγκρίνεται πρώτα από ανεξάρτητη αρχή στην Ευρώπη. Η δική σας υπηρεσία με ποιον τρόπο ενεπλάκησε όλη αυτή τη ε, διαδικασία. Είχατε κάνει παρατηρήσεις, είχατε δει. Δεν είναι δυνατόν να σας ελέγχει και εσάς η Boeing. Θα ήταν σαν ε, ε, η, να, να βάζουμε τη Volkswagen να ελέγχει τα ίδια της τα τα, οχήματα και όχι ανεξάρτητες αρχές. Τέλος, υπάρχει ανταγωνισμός και εντός της, αεροπορία, της αεροπλοείας, αλλά ε, υπάρχει και ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων ε, τρόπων μεταφοράς. Και το ζητούμενο και κριτήριο είναι πάντοτε η χαμηλή τιμή. Ναι, αλλά αν πάντοτε είναι το κριτήριο η χαμηλή τιμή, ίσως θα έπρεπε εμείς από την πλευρά μας να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες επενδύσεις για, να, για να ενισχυθεί ακριβώς αυτή η διάσταση της ασφάλειας. Διότι η ασφάλεια και η χαμηλότερη τιμή είναι δύο μεγέθη τα οποία δεν συμβαδίζουν πάντοτε. Εσάς σε ποιο βαθμό σας έχει επηρεάσει αυτή η προβληματική. Τέλος, Φυσικά η αίτηση θα είναι από την Boeing. Όταν θα ολοκληρωθεί η συζήτηση θέλουν να ξαναλάβουν έγκριση για τα αεροσκάφη τους. Εσείς τι θα κάνετε όμως. Πώς θα εξασφαλίσετε την ανεξαρτησία σας. Θα πείτε στους Αμερικάνους ότι θα ξαναπάρετε έγκριση μόνο αν αποκαταστήσετε τους κανόνες του 2005. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε έγκριση για να πούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μας υπαγορεύσει εμά η Boeing τι είναι, ποια θα είναι τα πρότυπα ασφαλεία στην Ευρώπη. Ερώτημα, ερώτημα προς εσάς, τι θα κάνετε. Ευχαριστώ κύριο Κράμερ, κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις έχω. Καταρχήν, εγώ θεωρώ συγχυστικό ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα και αυτό απλώς επιδεινώνει την κατάσταση ό,τι αφορά τη διαφάνεια του κατασκευαστή. Σε σχέση τώρα με τις τρεις ερωτήσει, καθώ είναι πολύ τεχνικά ζητήματα, θα ήθελα κάποιε διευκρινήσει. Από όσο γνωρίζετε, από πότε αυτά τα προβλήματα Φυσικά αφήνουμε ανοιχτή την έρευνα και δεν θα καταλήξουμε σε βιαστικά συμπεράσματα, αλλά ε, υπάρχει ένα θέμα αεροσκαφών. Κατά πόσο αφορά αυτό του τύπου τα αεροσκάφη του 737 MAX 8 ή αφορά και τα άλλα μοντέλα του 737. Η δεύτερη ερώτηση είναι, μπορούσαμε να γνωρίζουμε αν οι πιλότοι που χρησιμοποιούν αυτό το αεροσκάφος έχουν ε, πράγματι καταρτιστεί κατάλληλα και αν εσείς έχετε την δυνατότητα να καταλάβετε ε, με το αν ε, μπορεί να παρέμβει κάποιος ε, χειρονακτικά. Δηλαδή, ακούσα, ότι μπορούν να απενεργοποιηθούν αυτοί οι μηχανισμοί, όμως δεν ξέρω τι γίνεται με τους χρόνους. Ποιος καθόρισε τους χρόνους και τρίτον, ποιο είναι το πρωτόκολλο που ακολουθεί η ΆΣΑ για να μπορεί να αποφασίσει την αναστολή την ακύρωση των πτήσεων. Υπάρχουν κάποια κριτήρια ή είναι υποκειμενικό το θέμα. Τώρα το αυτό γιατί κάποιες εθνικές αρχές ε, προληπτικά έδρασαν και στις 7 το βράδυ ευρωπαϊκής ώρας ε, πήρατε εσείς την απόφαση όταν ήδη κάποιες εθνικές αρχές είχαν αποφασίσει σχετικά νωρίτερα. Σας ευχαριστούμε κυρία και κυρία Βάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Κύ, για την παρουσίασή σας. Εγώ έχω διαφορετικά ερωτήματα να σας θέσω, το οποίο επίσης θεωρώ ότι είναι ουσιώδη. Είχαμε στο παρελθόν το φαινόμενο μια, ένα καινοτόμο, μια καινοτόμα μηχανή, η Concord συγκεκριμένα, να μην καταφέρει τελικά να μπορεί να πετάει. Ε, παρόλο που ήταν ε, καινοτόμια, όπως είπα, η τεχνολογία που ε, ήταν ενταγμένη στα Concord. Για μένα το ερώτημα είναι, οι πιλότοι δεν θα πρέπει να καταρτίζονται και γύρω από ηλεκτρονικές τεχνολογίες για να μπορούν ακριβώς να είναι κυρίαρχοι των συστημάτων τα οποία καλούνται να χειρίζονται. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επανακαταρτίζονται διαρκώς οι, πολι... οι πιλότοι. Πώς μπορεί η ΕΑΣΑ να εξασφαλίσει, να εγγυηθεί ότι εκείνοι που θα κάνουν τις, ε, τους ελέγχους και τις εγκρίσεις ε, θα είναι ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Μπορεί να ακούγεται λίγο οξύμορο, αλλά όσο προχωράει η τεχνολογική πρόοδος, και φυσικά ούτε μπορούμε να φανταστούμε μεθαύριο, αύριο μεθαύριο τι θα έχουμε, ε, τι τεχνολογίες θα έχουμε, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι ελεγκτές, εκείνοι που δίνουν τις εγκρίσεις, είναι ενήμεροι. Ευχαριστώ κύριο Μπάρ. Ευχαριστώ κύριε Κι για, για την παρουσίασή σας. Έχω και εγώ δύο συγκεκριμένα ερωτήματα για την κατάρτιση. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την παρουσίασή σας για την προσωμείωση πτήσεων. Εντάσσονται ε, τέτοιες προσωμιώσεις στην εκπαίδευση των ε, πιλότων. Ε, εκπαιδεύονται για καταστάσεις εκτακτής ανάγκης, επικίνδυνες καταστάσεις. Αναφερθήκατε στην κατάρτιση, αλλά δεν ξέρω αν κατάλαβα αυτό που είπατε. Δεύτερο ερώτημα. Αυτό το MCAS είπατε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία του, του, κινητή, του, του, του όλου μηχανήματος, του όλου αεροσκάφους. Μπορεί ε, ένα αεροσκάφος πλέον να πλοηγηθεί, να πετάξει και χωρίς αυτό το δομικό στοιχείο. Ε, Ήθελα και εγώ να θέσω ένα ερώτημα. Ε, ε, είναι λίγο περίπλοκο βέβαια. Λοιπόν, γίνεται ένα πρώτο ατύχημα, έτσι, ένα πρώτο δυστύχημα πριν από μερικούς μήνες. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν λαμβάνει η χώρα μια έρευνα και οι υπηρεσίες οι διάφορες μεταξύ των οποίων η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κάνουν την έρευνά τους φαντάζομαι και εσείς ασχοληθήκατε με αυτό κατόπιν τούτου αν κατάλαβα καλά ο κατασκευαστής δίνει κάποιες ενδείξεις Κάποιε οδηγίε αν θέλετε, κατευθυντήριες γραμμέ προ του πιλότους. Είναι λίγο περίεργο αυτό, έτσι. Πρώτον, ο κατασκευαστή, έτσι. Ο κατασκευαστή το κάνει αυτό, όχι η υπηρεσία. Η Αμερικανική υπηρεσία δεν έχει φτάσει στην περάσματα ακόμα για το πρώτο ατύχημα, όπω ξέρουμε. Δεύτερον, εάν ο κατασκευαστή δίνει συστάσεις, συγκεκριμένες συστάσεις στους πιλότε, στους πιλότους, θα πει ότι έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποια ανομαλία ή κάτι που εν πάση διακυβεύει το αεροσκάφος. Η απάντηση λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, ότι ξέρετε τότε θα πρέπει να περάσετε, να περάσετε σε χειροκίνητο, σε χειροκίνητη πλοήγηση, ε, είναι, μια αρκετή. Είναι μια απάντηση για οτιδήποτε τελικά μπορεί να σημαίνει σε ένα αεροσκάφο. Τρίτον, πώς γίνεται ο ο κατασκευαστή που γνωρίζει τα πράγματα βέβαια, αλλά δεν είναι επιφορτισμένο με την έρευνα, να προτείνει μέτρα τροποποίησης, που σημαίνει ότι γνωρίζει κάποια πράγματα. Προτείνει λοιπόν λύσει. Και επ' αυτού εκείνη τη στιγμή, δηλαδή στι 6, 7, 8 Νοεμβρίου, η Αμερικανική υπηρεσία δεν παίρνει θέση. Δεν λέει τη γνώμη τη. Δεν επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο κατασκευαστή. Ούτε τον επικρίνει. Έχουμε λοιπόν την εντύπωση σε αυτή την υπόθεση, αν κατάλαβα καλά, υπάρχει ένα πρόβλημα με το σύστημα ψηφιακής διαχείρισης και ο κατασκευαστής ε, πιστεί την προσοχή στο πλήρωμα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι. Και λέει στην περίπτωση αυτή, ε, τα βγάζετε από την πρίζα όλα αυτά και κάνετε χειροκίνητη πλοήγηση. Ε, αντί να πει, ξέρετε, αφήνω το αεροπλάνο, το στο έδαφος διότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο οδήγησε σε 150 νεκρού, λέει αυτό. Ε, είναι πραγματικά απίστευτο, έτσι. Από τη στιγμή που το, η Boeing έδωσε νέες συστάσεις ε, προς τους πιλότους, δεν σημαίνει ότι έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει κάποιο θέμα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό όταν συμβαίνει κάτι, όταν, όταν προκύπτει. Εγώ δεν είμαι ειδικό στο θέμα αυτό. Όμως η σιωπή τη Αμερικανικής υπηρεσίας, το γεγονός ότι έκανε συστάσει ίδια η Boeing για πρώτο, το πρώτο ατύχημα και ότι παρόλα αυτά αυτό δεν μας οδήγησε να αποτρέψουμε ε, το δεύτερο, Μήπω τελικά δεν, αυτή η υπόθεση είναι πραγματικά εξαιρετικά σοβαρή ε, και σε νομικό επίπεδο. Δηλαδή ο κατασκευαστής αναγνώρισε κάτι και πρότεινε κάτι και αυτό δεν απέτρεψε το δεύτερο ατύχημα, οπότε είναι προφανές ότι έχει ευθύνη, αφού έγινε δεύτερο ατύχημα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, έτσι. Και το τελευταίο ερώτημα. Η ΕΑΣΑ όποια και είναι η θέση της Αμερικανικής ε, υπηρεσίας, ομοσπονδιακής υπηρεσίας, θα υποβάλει ε, την άδεια ε, πτήσης για αυτά τα, ε, για αυτά τα αεροπλάνα ε, στη δική σας σύμφωνη γνώμη. Λοιπόν, έχετε νομίζω πολλά να πας στα οποία πρέπει να απαντήσετε. Σας ακούμε με προσοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περάσω και πάλι στα αγγλικά διότι δεν γνωρίζω τους όρους στα γαλλικά. Και ξεκινάμε με τον κύριο Βαντενκάμπ. Ναι, όντω είναι στον τύπο αυτό. Δεν σας δίνω εδώ εμπιστευτικές πληροφορίες. Τα μαύρα κουτιά όντως εστάλησαν στο Παρίσι. Δεν είναι και πολλές οι χώρες στον κόσμο που έχουν τεχνικές δυνατότητες να επεξεργαστούν αυτά τα μαύρα κουτιά και η Γαλλία είναι μία από αυτές τις χώρες. Στο Παρίσι λοιπόν αυτά τα μαύρα κουτιά α, αναλύθηκαν χωρίς όμως ερμηνεία των δεδομένων. Δηλαδή η σχετική υπηρεσία έρευνας η γαλλική απλά ε, έχει βγάλει αυτά τα δεδομένα από τα μαύρα κουτιά και τα παίστηλε ε, στις αρχές της Αιθιοπίας. Και αυτό δείχνει ότι η αρχή έρευνα της Αιθιοπίας θέλει να έχει ένα πολύ κλειστό κύκλο γύρω από αυτήν την έρευνα. Να κάνει δηλαδή ό,τι μπορεί να κάνει εκεί, στην αντί Αμπέμπα, με την Αμερικανική, τις αρχές βέβαια, διότι από εκεί προέρχεται το αεροσκάφος. Θέλει όμως να περιορίσει οπωσδήποτε τους εμπλεκόμενους στην έρευνα. Όταν είπα ότι ζητήσαμε να συμμετάσχουμε στην έρευνα αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επίτροπος το ζήτησαν αυτό από τους συναδέλφους τους διότι σε μια, στο σχετικό κανονισμό για την έρευνα ατυχημάτων, διερεύνηση ατυχημάτων προβλέπεται ότι η χώρα που διενεργεί την έρευνα μπορεί να προσκαλέσει όποιον θέλει για να συμμετάσχει σε αυτή τη διερεύνηση. Βεβαίως κάποιες χώρες έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν μεταξύ των οποίων και η χώρα κατασκευή του αεροσκάφου και η χώρα βεβαίω ε, τη εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή οι αιθιοπικές αρχές θέλησαν ε, ε, θα μπορούσαν να μας καλέσουν εφόσον επιθυμούσαν ως παρατηρητές. Αυτό ζήτησε και ο Επίτροπος Μπούλτς τη Δευτέρα από την ομόλογο, ομόλογο της από την Αιθιοπία και αναμένουμε ακόμα την απάντηση. Η ΕΑΣΑ, σύμφωνα με τον κανονισμό 2.16 ε, για την διερεύνηση ατυχημάτων, όταν η αρχή ενός κράτους μέλους εμπλέκεται ως πιστοποιημένος εκπρόσωπος σε μία ε, έρευνα, τέτοιου είδους έρευνα, τότε πρέπει να συμμετάσχει και η ΆΣΑ ως τεχνικό σύμβουλος. Στην περίπτωση λοιπόν του downloading των δεδομένων, των στοιχείων του μαύρου κουτιών ήμασταν, ήμασταν παρόντε, ήμασταν εκεί. Δεν μπορούσαμε να συμμετάσχουμε στην επεξεργασία, δεν, δεν έλαβε χώρα επεξεργασία. Άρα μα κάλεσε η γαλλική υπηρεσία. Και αυτό πήγε καλά. Τώρα βέβαια εμείς ελπίζουμε ότι η αιθιοπική κυβέρνηση θα μας επιτρέψει να είμαστε παρατηρητές σε αυτή την έρευνα να γνωρίζουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα αν πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο σε ό,τι αφορά το Boeing 737 MAX. Για το δεύτερο ερώτημά σας τώρα κύριε Βεντενκάμπ για το επιχειρησιακό αυτό δελτίο της Bullet, της Boeing. Ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να επανέλθουμε στην παρουσίασή μου στο PowerPoint. Ε, αναφέρεται αυτό σε μία από τις ε, διαφάνειες, ε, εν πάση περιπτώσει, είναι μία σελίδα. Μία σελίδα. Δεν είναι και τόσο περίπλοκο. Ακόμα και εγώ μπορούσα να το καταλάβω. Είναι αρκετά κατανοητό. 6 Νοεμβρίου το δημοσίευσε αυτό η Boeing και η FAA δημοσίευσε την αντίστοιχη, το αντίστοιχο κείμενο στις 7 την επόμενη μέρα. 7 Νοεμβρίου. Τι λέμε λοιπόν εδώ, ότι όταν έχουν, εμφανίζονται μια σειρά από συμπτώματα και μάλιστα λέγεται πια τα συμπτώματα, υπάρχει ένα κατάλογος, τότε είναι πιο κάτω, είναι πιο κάτω. Εδώ, ναι. Μια σελίδα είναι έτσι. Εντάξει, βέβαια είναι μικρή χαρακτήρα για να το διαβάσετε εκεί, αλλά τι λέμε εδώ, αν εμφανιστεί κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, τότε πρέπει να κόψετε αυτή τη λειτουργία, να, την, να διακόψετε τη λειτουργία της, αυτή της εφαρμογής. Είναι απλό. Και έρχομαι στο ερώτημα του κυρίου Μπάρ και στο δικό σας ερώτημα και άλλα ερωτήματα που έθεσαν ε, ευρωβουλευτές. Έχετε απόλυτο δίκιο που το συνδέεται όλα αυτά με την κατάρτιση. Διότι αυτό που συνέβη ε, εντάξει, στο, στο δυστύχημα της Lion Air γνωρίζαμε, είπαμε προς τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, μας λένε ότι στην περίπτωση αυτή έχουμε ένα σένσορα AOA που δεν δίνει τις κατάλληλες πληροφορίες το σύστημα MCAS θα δώσει την οδηγία για βουτιά. Και θα δημιουργήσει βεβαίως μια επικίνδυνη κατάσταση. Εάν όμως το γνωρίζει αυτός, εφόσον κλείσει το σύστημα, μπορεί να συνεχίσει να πετάει. Στην περίπτωση λοιπόν της πτήσης Lion Air, υπήρχε ήδη ένα πρόβλημα στην προηγούμενη πτήση με τους sensors AOA και το πλήρωμα τότε είχε τη σωστή αντίδραση, το έκλεισε το σύστημα και προχώρησε. Βεβαίω είναι πάντα πιο εύκολο το λέει κανεί εκ των υστέρων. Έτσι πρέπει να είχαμε κάνει το τάδε και το δίνα. Όμω από πλευρά διαδικασία δεν είναι και τόσο περίπλοκο. Για να επανέλθω τώρα σε αυτό που είπε ο κ. Μπάρα. Όταν η Boeing και η FAA εξέδωσαν αυτά τα ανακοινωθέντα, αυτές τις οδηγίες, ότι αυτό θα ήταν εύκολο να εφαρμοστεί για το πλήρωμα. Και όντως, όταν το τσεκάραμε, όλα τα πληρώματα είχαν λάβει την πληροφορία αυτή και γνώριζαν, το γνώριζαν αυτό που βλέπετε εκεί. Τώρα αυτό που είναι αληθές και είναι θέμα ανθρώπινου παράγοντα, ερχόμαστε εδώ σε ένα από αυτά τα θέματα που έδωσε η κυρία Μάισνερ, η συμπεριφορά οποιοδήποτε ανθρώπινου όντω που σε μια πραγματική κατάσταση αντιμετωπίζει ε, ένα, μια συνθήκη όπου ε, χτυπάνε διάφορα καμπανάκια στον αγερμού, ε, τότε η συμπεριφορά του αλλάζει. Λοιπόν, στη Λάιονέρ, την προηγούμενη ακριβώ πτήση το πλήρωμα έκλεισε το σύστημα. Την, την επόμενη φορά δεν είχαν την, τη σωστή αντίδραση. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη τώρα στην περίπτωση της ε, Ethiopian Airlines, αλλά είναι πιθανό εκείνη τη στιγμή να μην σκέφτηκαν τα συγκεκριμένα, συγκεκριμένες οδηγίες ε, αυτού του bulletin, το οποίο δεν είναι ότι καλύτερο βέβαια, όντως διότι λέγεται, λέει ότι αν δείτε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σύμπτωμα, κλείστε το σύστημα. Ένα τέτοιο σύμπτωμα, κλείστε το σύστημα. Ε, το οποίο είναι κάτι απλό. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Εάν γνώρισαν τι ακριβώς συνέβαινε, δεν θα έκαναν αυτό που έκαναν, και δεν θα είχαμε το ατύχημα. Και ερχόμαστε σε κάτι που είπαν πολλοί από εσά. Εξετάσαμε τη βάση δεδομένων με, τα, με τις εκθέσεις. Από πληρώματα, ε, τις αναφορές, τις διάφορες, από τον κατασκευαστή, από τις αεροπορικές εταιρείε. Και στη βάση δεδομένων μας, δεν είναι παγκόσμια βέβαια η βάση δεδομένων μας, δεν είδαμε άλλα παραδείγματα παρεφερών ατυχημάτων. ...376 αεροσκάφη MAX ε, κυκλοφορούν παγκοσμίω, 50 περίπου στην Ευρώπη, εντάξει δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, στη βάση δεδομένων μας πάντων δεν είδαμε οποιοδήποτε στοιχείο που να δείχνει ότι είχαμε κάτι το παρεμφερές, κάτι, κάτι τέτοιο. Το κυρομελετήσαμε βέβαια μετά το, το, το δυστύχημα τη Lion Air. Εξετάσαμε ποιος είναι, ποια είναι η πιθανή αιτία του δυστυχήματος, πόσες φορές ε, έχουμε δει να συμβαίνει κάτι τέτοιο, μηδέν, και βεβαίω εξετάσαμε τι πρότεινε η Boeing και η FAA να ενημερωθούν και να καταρτιστούν τα μέλη του πληρώματος έτσι ώστε αν ξανασυμβεί αυτό να, πρέπει, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, να κλείσουν δηλαδή το σύστημα και βεβαίω εκ των υστέρων ε, ενδεχομένω να είχαμε κάνει κάτι άλλο αλλά τότε θεωρήσαμε ότι ήταν μια καλή, μια αποδεκτή ένα αποδεκτό μέτρο ασφάλειας αναμένοντας την επικαιροποίηση του, λογισμικού το οποίο προετοιμάζει Boeing. που εξετάζει το MCAS εξασφαλίζει ότι μπορεί κανείς δηλαδή, να, μπορεί να κλείνει πιο εύκολα ή εν να μην από, να μην, ε, από μόνο του, να μην αντιδράει με έναν τρόπο μόνο και μόνο επειδή δύο σένσορες στέλνουν μια πληροφορία και εξετάζεται βεβαίω τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε δύο σένσορες που δίνουν ε, αντικρουόμενες πληροφορίες. Διότι είναι κάτι που στην περίπτωση στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Κράμερ προηγουμένως για, το, για την Airbus υπάρχουν τρεις σένσορες και αν ένας δεν λειτουργήσει υπάρχουν δύο ακόμα. Εάν, υπάρχει, αν υπάρχουν δεκρόμενες πληροφορίες μεταξύ των δύο και του ενός σένσορ υπάρχει ένας μηχανισμός ε, το οποίο το επιλύει αυτό, ε, είναι διαφορετική η δομή. Αυτά είναι, αυτές, είναι, λοιπόν οι ενημερώσεις επικαιροποίησης του λογισμικού για τους σένσορες. Θέλω να σας ε, πω, διότι ελέγχεται σε πολλές παρεμβάσεις, Αυτές οι επικαιροποιήσεις του λογισμικού εμείς θα τις εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Και θα πάμε και πίσω και στη δομή του ΕΜΚΑΣ να δούμε όλα τα ζητήματα αυτά και πώς το Boeing τα διαχειρίζεται. Και από την πλευρά μας δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να πετάξει το αεροσκάφος εάν δεν βρούμε αποδεκτές απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Ό,τι και αν κάνει η FAA. Ό,τι και αν κάνει η FAA. Αυτή είναι μια εγγύηση που αναλαμβάνω εγώ εδώ προσωπικά μπροστά σας. Μια δέσμευση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαδικασία για την απαγόρευση πτήσης. Απαγόρευση απογείωσης. Κάποια μέλη της Ένωσης όντως αποφάσισαν να απαγορεύσουν ε, ε να απαγορεύσουν να, να, να απογειωθεί, να απαγορεύσουν την χρήση του εναέριου χώρου. Έτσι. Ε, κάποιοι το κάνουν μερικές ώρες πριν. Γιατί εμείς αργήσαμε λίγο. Πρώτον, διότι Κάναμε πολλές, πραγματικά πολλές τεχνικές αναλύσεις για να φτάσουμε σε αυτή την απόφαση. Είχαμε πολλές συζητήσεις σε εσωτερικό επίπεδο με τα διάφορα πάνελ εμπειρογνωμόνων. Εξετάσαμε τους διάφορους λόγους για το ατύχημα, για το δυστύχημα αυτό. Σας, θυμάμαι, σας θυμίζω ότι δεν συμμετείχαμε στην έρευνα, έτσι. Οπότε είχαμε λίγες πληροφορίες στη διάθεσή μας. Όμως όλοι οι εμπειρογνώμονές μας ασχολιόταν με τα Boeing και τα, Air, Airbus ε, για να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι για αυτό το ατύχημα, ποια είναι, ε, ποιες οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας και ποια είναι η απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Την Τρίτη το πρωί λάβαμε μια ενημέρωση η DSB λέει, δηλαδή, που βασίζεται στο δορυφόρο από τις Ιρλανδικές αρχές που είναι ένας πάροχος η DSB παγκοσμίω. Ε, με βάση τις πληροφορίες αυτές μπορέσαμε να εξεργαστούμε ε, έτσι και να εξετάσουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ε, τροχιά του αεροσκάφους κτλ. Πολλές άλλες χώρες δεν έχουν την πληροφορία αυτή. Τέλος, αυτό που θέλησαμε να κάνουμε ήταν να ενημερώσουμε, να επικοινωνήσουμε, να συζητήσουμε με τους αδέλφους μας ε, της FAA για την απόφαση που παίρναμε. Όπως ξέρετε υπάρχει μια διαφορά 6-7 ωρών με τις ΗΠΑ και μας πήρε περισσότερο χρόνο. Η Βρετανία αποφάσισε στις 12, 1 και εμείς στις 5. τέθηκε ένα ζήτημα, ένα ερώτημα για τους διάφορους τύπους ε, σένσορων. Δεν γνωρίζω αν κάποιοι σένσορες είναι πιο ακριβοί ή πιο φτηνοί. Εγώ πως ένας είναι ο τύπος από όσο ξέρω που χρησιμοποιείται και δεν έχω ακούσει τίποτα για πιο φθηνούς και πιο ακριβούς σένσορες. Ξέρετε, το κόστος ενός σένσορα σε σχέση με το κόστος του αεροσκάφους είναι πολύ περιορισμένο. Ναι, πάντως υπήρξαν εκθέσεις αρκετά πιστικές ότι το, το αεροσκάφος του, των Ethiopian Airlines αλλά και το, της Lion Air είχαν μια λειτου, συγκεκριμένη λειτουργία των σένσορων AOA που είναι το βασικό μοντέλο και αν κάποιος είχε δαπανίσει περισσότερα χρήματα υπήρχε ένα άλλο, μια, άλλη, μια άλλη εκδοχή, ένα άλλο μοντέλο. Ε, δεν ξέρω αν έχει σχέση αυτό να κάνει με το Max 8 ή το Max 9. Πάντως ε, υπάρχουν σίγουρα διαφορές ε, σε ό,τι αφορά το τι επιλέγουν οι αεροπορικέ εταιρείε να παραγγείλουν. There is one thing which... Υπάρχει κάτι που δεν συνδέεται με τους σένσορες, ε, είναι ένα display στο cockpit, πως παρουσιάζονται οι πληροφορίες για το αν συμφωνούν ή όχι οι αισθητήρε και αυτό είναι μέρος της αλλαγής του λογισμικού. Αυτό θα γίνεται ε, ουσιαστικά προγραμματισμένο, γιατί πριν ε, ήταν ε, επιλογή. Θα γίνεται δηλαδή το άλλος. Υπήρξαν και κάποια σχόλια. Νομίζω από την κυρία Ντεμόντε για το θέμα της κατάρτισης. τουλάχιστον είναι κάτι που αφορά από το 737 ε, και τις άλλες εκδοχές του 737 το MCAS υπάρχει μόνο στο MAX. Έτσι λοιπόν δεν ε, υπάρχει σε άλλες εκδοχές του 737 και συγκεκριμένα στην γενιά ή στην ε, προηγούμενη γενιά στο 737. Ένα από τα κυρία χαρακτηριστικά της οικογένειας του 737 είναι αυτό που αποκαλούμε ικανότητα κατάρτισης ε, προς τα πάνω. Δηλαδή αν έχεις μία άδεια να πιλοτάρεις ένα 737 τότε με ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή παραπάνω κατάρτιση μπορείς να πετάξεις ε, ένα F37 Max ή ένα F37 παλιότερης γενιάς. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των αδειών Boeing, κυρίως για το F37. Εμείς θα τα εξετάσουμε όλα αυτά πάρα πολύ λεπτομερός και θα επανέλθουμε σε πάρα πολλά από τα σχόλια που κάνατε. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ε, η αναβάθμιση του λογισμικού που θα προταθεί από την Boeing δεν θα είναι ασφαλής μόνο σε ό,τι αφορά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την έγκριση, αλλά θα συνοδεύεται επίσης και από τις κατάλληλες απαιτήσει κατάρτισης και τις εξελίξεις για την κατάρτιση που θα είναι απαραίτητε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πιλότοι όχι μόνο θα λάβουν αυτές τις πληροφορίες, αλλά θα είναι και καταρτισμένοι, προκειμένου αυτόματα να μπορούν να κάνουν ό,τι απαιτείται από αυτούς, να αντιμετωπίζουν ε, μια προβληματική κατάσταση. Λοιπόν, ο κατασκευαστής ε, είδε ότι το σύστημά του θα μπορούσε να είναι ελαττωματικό. Το είδε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είδε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στο θάνατο 157 ανθρώπων σε μια συντριβή. Τρίτον, ε, αντίδρασε και είπε «Αχ, κόψτε το! Έτσι θα πάει καλύτερα». Ε, Παραδείγματο χάρη, όταν ένα κατασκευαστή αυτοκινήτων ε, βλέπει ότι ε, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον έλεγχο τη ταχύτητα, αποσύρει το όχημα. Όμω εδώ, στην περίπτωση αυτή, άφησαν να πετάνε τεροσκάφη με ένα σύστημα που μπορεί να θεωρεί το προβληματικό. Και εντάξει, ένα κινητήρα μπορεί να πάρει φωτιά, εντάξει, δεν είναι πολύπλοκο, κόψτε το. Ε, συμβαίνουν αυτά. Δεν χρειάζεται ε, να τα ρίχνουμε στο Κοιτάξτε τώρα, είναι κάπως ε, τρελό όλο αυτό. Εγώ αναφέρω εδώ ποιος ε, έχει την ενοχή. Κυρίως όταν αλλάζει ένα σύστημα αλλά οι πιλότοι δεν ενημερώνονται για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται από εδώ και στο εξή. Είναι σαφές ποιος είναι, ευθύ, ε, ποιος είναι υπεύθυνος δεν υπάρχει ποινή, δεν υπάρχει κύρωση πρόστιμο και μάλιστα υψηλό, γιατί ακριβώς έγινε μια αλλαγή και δεν ενημερώθηκαν οι πιλότοι για το τι πρέπει να κάνουν αν συμβεί το ένα ή το άλλο. Είναι απίθανο αυτό που έχουμε εδώ μπροστά μας. Βιμ. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις και τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Όμως, πραγματικά αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι η λειτουργία του συμπιλότου. Όταν απαντήσετε στον κύριο Μπάχ, είπατε ότι μπορεί οι άνθρωποι να συμπεριφερθούν διαφορετικά όταν είναι σε μια αίθουσα ή όταν είναι σε πραγματικές συνθήκες, στην πραγματική ζωή. Αλλά συνήθως νομίζω ότι ο έτερος πιλότος δεν διαβάζει περιοδικά βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει τον πιλότο. Ισμαήλ. Ευχαριστώ. Δεν άκουσα απάντηση στο ερώτημά μου. Είχαμε το, το δυστύχημα του Νοεμβρίου του 2019. Είναι πλέον Μάρτιος του 18. Είναι πλέον Μάρτιος του 19. Αν κατάλαβα σωστά, είπατε ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε η Boeing με την αναβάθμιση του λογισμικού σας φάνηκε επαρκής. Η απάντηση που έδωσε η Boeing είπατε ότι θεωρήσατε ότι ήταν επαρκής με αυτή την αναβάθμιση του λογισμικού στην οποία προέβη. Αλήθεια το είπατε αυτό. Και εσάς τι σας έκανε να πιστεύετε ότι μια αναβάθμιση του λογισμικού θα μπορούσε να επιλύσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα ή θα μπορούσε να εμποδίσει ε, την επανεμφάνιση, μια πιθανή επανεμφάνιση αυτού του φαινομένου. Και ξέρετε, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό, διότι τα, οι διάφορες, τα, τα, διάφορα πειράγματα στα λογισμικά τα έχουμε δει και στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και ξέρετε ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο να λύνονται μέσω του, του software τα προβλήματα. Ο κύριος Κράμερ, ένα πολύ σύντομο ερώτημα. Το λογισμικό ήταν αναγκαίο γιατί η Boeing βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την Airbus και ήθελε να είναι όσο καλή ήταν και η Airbus. Γι' αυτό λοιπόν το να κατασκευάσουν ένα νέο από την αρχή, ένα νέο μοντέλο ε, ήταν πάρα θα ήταν πολύ χρονοβόρο οπότε επέλεξαν να αλλάξουν απλά τον παλιό τους κινητήρα αλλάζοντας κάποια δομικά στοιχεία, αλλάζοντας την ισορροπία την εσωτερική του αεροσκάφους ε, Κάτι που τελικά ήταν εκείνο που δημιούργησε τα προβλήματα γιατί ακριβώς το κέντρο βάρους του αεροσκάφους βρισκόταν πλέον στο, ε, σε ένα νέο σημείο, σε ένα διαφορετικό σημείο, κάτι το οποίο δεν το γνώριζαν οι πιλότοι. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν ο ανταγωνισμός, διότι επιχειρήθηκε από την Boeing να σταθεί στον ανταγωνισμό αλλάζοντα επιμέρου κάποια στοιχεία του παλιού του κινητήρα αντί να φτιάξουν έναν καινούριο. Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Πρέπει να απαντήσετε πάρα πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στον Πατρίκ για να ολοκληρώσει. Ξέρω ότι υπάρχουν έντονα συναισθήματα, αλλά νομίζω ότι δόθηκαν πολύ συγκεκριμένε απαντήσει στι ερωτήσει. Μάλιστα, κυρία Ντεμόντε, ευχαριστώ. Ήταν σύντομη συνάδελφα, αλλά θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στις ε, ερωτήσεις. Πραγματικά ανησυχεί πάρα πολύ η κοινωνία. Εγώ δώσα μια συνέντευξη σε ένα εθνικό ραδιόφωνο και μου ζήτησαν να δώσω απαντήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να μας δώσετε εσείς ε, πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις σε σχέση με την ε, συμβατότητα της άδειας. Αυτό τι σημαίνει ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να αφορά και άλλα μοντέλα του 737 ή όχι, αφορά μόνο το MAX 8. Η δεύτερη ερώτηση ήταν, είμαστε βέβαιοι και ποιος μας διαβεβαιώνει ότι αρκεί ο χρόνος για να παρέμβει κάποιος χειρονακτικά. Και τρίτη ερώτηση, έχετε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που μας δείχνει πώς μπορεί να παρέμβει κάποιος όταν υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό, μέσα σε ποιο χρόνο πρέπει να αντιδράσει κτλ. Um, <coughs> θα ήθελα να συνεχίσετε τις ερωτήσεις σας ε, και να μπορέσω να φύγω από την αίθουσα γιατί θα είχε τελειώσει ο χρόνος, όμως δυστυχώς δεν με άφησε ο πρόεδρος. Ναι, αναφερθήκατε σε διάφορα θέματα. Να απαντήσω στον κύριο Κράμερ καταρχήν. Νομίζω ότι είναι καλός ο ανταγωνισμός γενικός γενικά. Και είναι γεγονός ότι η Airbus ε, βασικά είχε την ε, οικογένεια 20 ε, και έβαλε μια, ένα νέο κινητήρα και είναι λογικό ότι προσπαθεί να βάλει ένα νέο κινητήρα και η Boeing στην οικογένεια 737. Είναι λογικό σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο. Τώρα, εδώ ε, που επισέρχεται αυτό το λογισμικό. Σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου έχουμε κάποιες ε, στροφές με υψηλή ταχύτητα, η ε, απώλεια στήριξη, η συμπεριφορά του 737 με τους νέους κινητήρες που ήταν πιο βαργοί, δεν είναι ακριβώς η ίδια όπως με τα άλλα 737. Και γι' αυτό στην έκκληση να είναι όσο δυνατόν πιο κοντά τα χαρακτηριστικά μεταξύ των διάφορων γενιών, η Boeing σχεδίασε αυτό το λογισμικό για να δώσει, την, να υδατηρήσει, συγγνώμη, την ίδια συμπεριφορά ε, στο αεροσκάφος Max, αν και είναι διαφορετικό το κέντρο βάρους και το κέντρο δράνειας. Βέβαια, μπορώ να γνωρίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. και δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική η κατάσταση. you again. Μπορώ και μόνο να σας υποσχεθώ εκ νέου ότι θα διερευνήσουμε εις βάθος οποιασδήποτε μελλοντικής πρότασης οποιαδήποτε μελλοντική πρόταση της Boeing και για να επανέλθω σας είπατε θα διασφαλίσουμε ότι όχι μόνο θα γίνει σωστά το τεχνικό μέρος της ανάπτυξης με την ανάλυση όλες τις αιτίε που προκαλούν αποτυχία λειτουργίας, αλλά θα διασφαλίσουμε ότι και η σχετική κατάρτιση να είναι υποχρεωτική για όλους τους πιλότους. Για να απαντήσω κάποια από τα σχόλιά σας. Το να έχουμε δύο πιλότους στο πλήρωμα είναι πολύ καλό ταυτόχρονα γιατί έχεις ουσιαστικά τέσσερα μάτια, αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι και κακό. Γιατί ξέρετε ότι οι πιλότοι ως αντανακλαστικά μπορούν να δώσουν ε, κάποιες ε, εντολές ε, αλληλοσυγκρόμενες στο αεροσκάφος. Μόνο ένας πιλότος κάθε φορά έχει την ε, δίκηση του αεροσκάφου ε, και ο άλλο τον βοηθά, αλλά ταυτόχρονα δεν πλοηγεί. Και στην ε, περίπτωση της Lion στο σκέλος της πτήσης πριν από το τύχημα μεταξύ των δύο πιλότων μπόρεσαν να βρουν μια λύση. Ενώ σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση αν επιβεβαιωθεί ότι αυτή ήταν πραγματική αιτία του δυστυχήματος δεν μπόρεσαν να βρουν λύση. Γι' αυτό τόσο πολλά εξαρτώνται από την κατάρτιση. Η κατάρτιση δεν αφορά μόνο του μονομένους πιλότους, αλλά και τους δύο πιλότους μαζί. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να δοκιμαστεί αυτό σε ένα περιβάλλον προσωμιωτή που να είναι το πιο κοντά σε πραγματικές συνθήκες. Για να υπάρχει και αυτή η εμπειρία, να λειτουργούν δηλαδή τα πληρώματα μαζί. Κύριε Πρόεδρε, τέλος. Οι πιλότοι δεν οδηγούν αυτοκίνητα, δεν οδηγεί αυτοκινήτων. Λαμβάνουν ιδιαίτερα ακριβέ καταρτήσεις. Είναι εμπειρογνώμονες στην, στο χειρισμό του αεροσκάφους και στο χειρισμό των συστημάτων ε, σε περιπτώσει όπου δεν λειτουργεί αυτόματα το αυτόματο σύστημα, γι' αυτό χρειαζόμαστε του πιλότους, διαφορετικά θα γινόνταν όλα αυτόματα. Αλλά σήμερα ο πιλότο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά ασφαλεία ε, του σχεδιασμού του αεροσκάφου. Και αυτό είναι ο λόγο, που σε ορισμένε περιπτώσει, δίνονται οδηγίες στους πιλότους για το πώς θα αντιμετωπίσουν κάτι που δεν λειτουργεί σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο. Δεν λέω ότι αυτό είναι δικαιολογία για την Boeing, αλλά αυτό εξηγεί τη διαφορά που υπάρχει σε διάφορους τομείς αεροπλοείας και τι συμβαίνει. Εντάξει. Είμαι σίγουρη ότι και διερμηνείς έχουν παθιαστεί με αυτό το θέμα, αλλά βέβαια έχει εξαντληθεί ο χρόνος μας. Ah bon, on peut continuer alors. Alors, euh, si ça n'est pas abusé, euh, et qu'on a encore un peu Μάλιστα, από τότε έχουμε λίγο ακόμα χρόνο. Ε, κανένα πρόβλημα. Απλά νόμιζα ότι δεν είχαμε χρόνο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πατρίκ, ε, κοιτάξτε. Σίγουρα οι πιλότοι δεν είναι οδηγοί αυτοκινήτων. Αλλά τέλο πάντων σε ένα αυτοκίνητο τέσσερα άτομα είμαστε, όχι 200. Λοιπόν, για να ξανάρθω στο θέμα τη ερώτηση Ερτούγκη για το λογισμικό, συγγνώμη δεν απάντησα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα ότι με ένα νέο είδο λογισμικού δεν λύνουμε απαραίτητο όλα τα ζητήματα. Αυτό που θέλουμε να λύσουμε είναι ε, όλες οι περιπτώσεις όπου έχουμε αποτυχία λειτουργίας του συστήματος. Αν έχετε ένα λογισμικό που κάνει κάτι και βλέπεις ότι σε ορισμένε περιπτώσεις δεν κάνει τη δουλειά του, απλώς διορθώνεις ε, αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό που Μπορεί να φαίνεται κάτι σαν ένα quick fix, σαν γρήγορη διόρθωση που προτείνεται από την Boeing στην ε, περίπτωση αυτή. Είχαν δηλαδή ένα πρόβλημα με το λογισμικό και το διορθώνουν. Αν απλώ κάνουμε αυτό, σύμφωνα απόλυτα μαζί σα ότι αυτό δεν αρκεί. Αλλά τι σκοπεύουμε εμεί να κάνουμε. Να φτάσουμε ει βάθο και να αναλύσουμε όλο το συνδυασμό όχι μόνο του software αλλά και τη αλληλεπίδραση μεταξύ του λογισμικού και των ε, διάφορων υλικών συστημάτων στο πιλωτήριο και επίσης ε, και την ε, διαπαφή ανθρώπου μηχανής. Δηλαδή όχι μόνο να δούμε τις αλλαγές του λογισμικού που είναι κάτι επιφανειακό, αλλά να δούμε και όσα κρύβονται από πίσω. Και όλη για την αρχιτεκτονική του συστήματος. Απαντά αυτή την ερώτησή σας. Ναι, αλλά ε, στο μεταξύ φαντάζομαι ότι όλοι όσοι έχουν ε, τέτοια αεροσκάφη δεν θα τους επιτρέπεται να, τα πετάνε. Συγγνώμη, για το διεθνές δίκαιο θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι. Γιατί είναι πιθανόν οι ΙΠΑ να έχουν παραβιάσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Για το διεθνές δίκαιο. Βάσει του διεθνούς δικαίου όλα τα αεροσκάφη που κινούνται στον εναέριο χώρο της, ε, των χωρών που είναι, που είναι καταχωρημένα στην, ε, στην Ευρώπη πρέπει να έχουν εγκριθεί από εμάς. Όπως είπα, στην περίπτωση της CFA έχουμε ε, διμερείς συμφωνίες οι οποίε μας επιτρέπουν να βασιζόμαστε εμεί σε και εκείνοι σε εμά. Και έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία μαζί τους. Όμως, έχει συμβεί να ε, διαφωνούμε στο παρελθόν. Προσπαθούμε, προσπαθούμε να μην φτάνουμε τα πράγματα σε αυτό το σημείο, αλλά ε, από άποψη διεθνούς δικαίου κάτι τέτοιο είναι πιθανό να διαφωνούν οι δύο υπηρεσίες. Γι' αυτό και σας είπα ότι εμείς σκοπεύουμε να εξετάσουμε σε βάθος τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Θα το κάνουμε. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό σε πλήρη και απόλυτο συντονισμό με τους συναδέλφους της CFAA, e Όμως εμείς, ανεξάρτητα από αυτό, θα κάνουμε τη δουλειά μας στο βαθμό που πρέπει, που θεωρούμε εμείς ότι πρέπει, για να έχουμε ασφαλή αεροσκάφη. Κύριε Ντεμόντε. Ευχαριστώ. Παίρνω για τρίτη φορά τον λόγο και ζητώ συγγνώμη. Δεν έχω όμως καταλάβει ακόμη αν το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ε, προβλήματα και σε άλλα μοντέλα του 737. Είμαστε σίγουροι ότι το πρόβλημα αυτό αφορά μόνο το MAX 8. Να το ξεκαθαρίσω. Το πρόβλημα που εντοπίσαμε στη Lion Air γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώ έγινε στι αιθιοπικέ γραμμές. Αν όμως είναι ε, το ίδιο πρόβλημα, αν ήταν η ίδια αιτία, αυτό αφορά μόνο το MAX, το 737 MAX. Τα παλιότερα μοντέλα δεν έχουν τα, τα ίδια συστήματα, δεν έχουν το ίδιο MCAS. Οπότε δεν τα αφορά, δεν κινδυνεύουν από το ίδιο πρόβλημα. Τελευταία ερώτηση κύριε Κράμερ. Αν η Boeing είχε αποφασίσει τότε να περιμένουμε καλύτερα 3-4 χρόνια να κατασκευάσουμε ένα νέο αεροσκάφος το οποίο θα είναι συγκρίσιμο με εκείνο της Airbus. Αν είχε γίνει αυτό, τότε μπορεί να είχαν μείνει λίγο πίσω στον ανταγωνισμό, αλλά θα είχαν αποφευθεί αυτά τα δύο ατυχήματα. Με συμφωνείτε μαζί μου σε αυτό? Uh, you know, if, if, ε, if αν η Boeing είχε αποφασίσει να κατασκευάσει ένα ολοκένουργιο αεροσκάφο, ίσως θα μπορούσαν να είχαν να αντιμετωπίσει και νέα διαφορετικά, διαφορετικού είδους προβλήματα. Δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Τα 737 είναι το αεροσκάφος που έχει πολιθεί περισσότερο από κάθε άλλο στον κόσμο. Έχει ιστορία 50 ετών και πάνω. Το να γίνουν αυτές κάποιες προσαρμογές στον ε, κινητήρα θεωρήθηκε ότι θα ήταν, ήταν προτιμότερη επιλογή. Ε, τώρα, το, γιατί δεν, κατε, δεν αποφάσισαν να κατασκευάσουν ένα αεροσκάφο είναι δική τη υπόθεση, δεν μπορώ να τη σχολιάσω εγώ. Θέλετε να πείτε κάτι ε, για να κλείσουμε. Ναι, εγώ θέλω απλώς να επαναλάβω ότι θα πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις για να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας. Θα είμαστε ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε πολιτική ή οικονομική πίεση που μπορεί να ασκηθεί επάνω μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Μάλιστα. Εμείς ευχαριστούμε το Γενικό Διευθυντή και τους συνεργάτες του. Διευθυντή πολύ ειλικρινή, έτσι, ανοιχτή συζήτηση και ελπίζουμε να μπορέσουμε να μας διαφωτίσετε για το θέμα αυτό, το οποίο και τις υποθέσεις που είχαν πάρα πολλά θύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη πρέπει ακόμα να πω στους συναδέλφους πριν φύγουν ότι τους δίνω ραντεβού για τις 8 Απριλίου επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.